Αγαπητοί συνάδελφοι, Καλώ ήλθατε. Έχει λάβει χώρα μια αλλαγή τη ημέρησιας διάταξη. Έλαβε χώρα μια έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών και γι' αυτό το λόγο πρέπει και εμεί να απασχοληθούμε με το θέμα τη Ουκρανίας. και υπάρχει ο εκπρόσωπος της Πεσβείας της Ουκρανίας καθώς και ο αρμόδιος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για την έγκριση της τροποποίησης αυτής. Δεν έχω να κάνω καθόλου ανακοινώσει. Ερχόμαστε τώρα στις ψηφοφορίες. Έχουμε μία γνωμοδότηση του κυρίου Έλα Θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια. Δεν χρειάζεται να σας καθυστερήσω, λέει κύριο Σέλε. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ε, κοινή ε, συζήτηση μεταξύ Επιτροπής ΣΕΔΕ και Επιτροπής Εξωτερικών Θεμάτων. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι ανάγκες χρηματοδότησης των εξωτερικών ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό οδήγησε σε επίπεδο σχεδόν παραλογισμού. Είχαμε πολλές καθυστερήσεις για την έναρξη επιχειρήσεων λόγω προβλημάτων αυτού του είδους. Κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητής. Γνωρίζετε ότι έχουμε προβλήματα όπως αυτό της Ουκρανίας. Κλείνει και πάλι ο ομιλητής το μικρόφωνο του. Έχουμε λοιπόν καθυστερήσει τη τάξη ε, του μισού ή ενό χρόνου και μετά στο πολιτικό κομμάτι μια επιχείρηση ξεχωρίζουν διάφορε δράσει οι οποίε έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και διαφορετικό καταλογισμό στον προπολογισμό. Για όλου αυτού του λόγου είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Ήταν σε επαφή και με τον ε, αρμόδιο τη Επιτροπής Προϋπολογισμών και έχουμε καταλήξει σε αυτή τη γνωμοδότηση η οποία έχει σαν στόχο να αλλάξει το σχεδιασμό σε δημοσιονομικό επίπεδο για τις ενέργειες αυτές πολιτικού χαρακτήρα τη εξωτερική πολιτικής επειδή της ε, εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο ο οποίο θέλει να λάβει το λόγο. Μπορούμε να ψηφίσουμε, λέει ο πρόεδρος Μπλοκ. Η υπέρ της 2. Κατά αποχές δεκτή. Εκπίπτει η τροπολογία ενός εκ τούτου και μπορούμε ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε το σύνολο της χρωμοδότησης. <coughs> Άρχεται η ψηφοφορία. Abstimmung ist geschlossen. Με δύο ε, αποχές, τρεις ψήφους κατά 64 ψήφους υπέρ, εγκρίνεται η γνωμοδότηση, συγχαίρω τον εισηγητή και η κυρία και επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είχε εγκριθεί αυτή η γνωμοδότηση. Wir 4. Περνάμε στο σημείο 4 τώρα. Προϋπολογισμός 2013. Απαλλαγή για τα θέματα Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε την κυρία Γέχτε Μάχη, η οποία είναι η εισηγήτρια. την οποία θα εκπροσωπήσει ο κ. Άουστε Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να αντικαταστήσω τη συνάδελφό μου την κυρία Γιάχτε Μάχη, η οποία δυστυχώ δεν ήταν σε θέση να είναι παρούσα στη σημερινή συνεδρίαση. η κυρία Γιάχτε Μάχη θα ήθελε να ευχαριστήσει του συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες για τη σημαντική του συνεισφορά στις δύο αυτές γνωμοδοτήσεις. Υποστηρίζει το μεγαλύτερο μέρο των τροπολογιών. Η Ανελή χαίρεται για το γεγονός ότι υπάρχει συναντήληψη μεταξύ των πολιτικών ομάδων για τα θέματα αυτά. Και δεύτερον, καλωσορίζει τη μείωση του ποσοστού ουσιαστικών σφαλμάτων το 2013 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις και κενά σε σχέση με τις δαπάνες της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα διαδικασία για ελέγχου για να αποφευθούν τέτοια σφάλματα στο μέλλον. Και επίσης ανησυχεί ιδιαίτερα για τις ε, καταγγελίες διαφθοράς για την EULEX στο κοσφοπέδιο. Και ελπίζω ότι θα μπορέσει να συμπληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν οι διαδικασίες έρευνα και να υπάρξει πλήρης πληροφόρηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή για την απάτη και την διαφθορά η Ανεργία Θεμάχη Επίσης χαιρετίζει το γεγονός ότι είναι ο, τρότος, ο τρίτος χρόνος ο τρίτο οικονομικό χρόνο, στον οποίο η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση εφάρμοσε τον προπολογισμό τη χωρί ουσιαστικά σφάλματα. Αλλά εκφράζει την ανησυχία τη για την έλλειψη ισορροπίας σε γεωγραφικό επίπεδο και επίπεδο φύλων σε ό,τι αφορά τι προσλήψει ε, στελεχών τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και θεωρεί ότι είναι υπέρβαρη στην κεφαλή η διοικητική δομή της υπηρεσίας εξωτερικής ε, δράσης και είναι μεγάλη η εξάρτηση από θέσεις υψηλού επίπεδου. Τονίζει η κυρία και επίση την θέληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενσωματωθεί ο ύπατο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να είναι καλύτερη η λειτουργία του προπολογισμού και θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνοχή τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Αυτά λοιπόν είναι το μήνυμα που θέλει να μας μεταφέρει η κυρία Μάχη. Χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την, την συγκήτρια κυρία Μάχη για τα σχέδιο το οποίο πολύ καλά έχει διατυπώσει και το οποίο λαμβάνει υπόψη τα κεντρικά σημεία. Θα ήθελα επίσης να επιμείνω όσον αφορά την απαλλαγή για τις, <coughs> την, ε, τους εκτελεστικούς οργανισμούς όσον αφορά τα υποθέσεις διαφθοράς. Τουλάχιστον όσον αφορά την Όλεξ Κωσυφοπέδη θα πρέπει να σεβαστούμε την αμεροληψία για την έρευνα που είναι υπό εξέλιξη και να μην ε, ε, υποχωρήσουμε σε πιέσεις ε, ακόμα. Ε, νομίζω πως όλα αυτά που αναφέρει η κυρία Γεχτερμάκη είναι εξαιρετικά χρήσιμα, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τον καλύτερο συντονισμό και την καλύτερη, ε, τη μεγαλύτερη ευελιξία για τη διαχείριση των κρίσεων. Όσον αφορά την ε, απαλλαγή για την ε, υπηρεσία εξωτερική δράση, Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε μια τροπολογία που αφορά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με τη δυσκολία των αντιπροσωπιών να διαχειριστούν τις προσφορές ε, για δημόσιους διαγωνισμούς ε, και είναι σημαντικό η αντιπροσωπεία να έχει αυτή τη στήριξη όχι μόνο για να τηρήσει καλύτερα τον δημοσιονομικό κανονισμό αλλά και έτσι ώστε οι επικεφαλή των αντιπροσωπιών να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην καρδιά της αποστολής τους, δηλαδή της εκπροσώπησης της Ένωσης. Όσον αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες δεν βρίσκω να υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες εκτός από την τροπολογία 6 που θεωρώ ότι είναι μια τροπολογία που είναι αντίθετη με μια θέση μάλλον που είναι κοντά στη θέση που θα υιοθετήσει το ΕΛΚ, αλλά ε, η συζητήσει είναι υπό εξέλιξη ακόμα. Οπότε να συγχαρώ ακόμη μια φορά για την εξαιρετική ε, εργασία την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια Σύμφωνο, καταρχήν σε πάρα πολλά σημεία με την γραμμοδότησή της. Βέβαια θα πρέπει εδώ να ληφθεί υπόψη η γενική μας στάση για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες κατά της EULEX στο Κόσοβο για διαφθορά, θα πρέπει, νομίζω ότι αφού έχουν γίνει απαραίτητες έρευνες, να αντλήσουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρξει και μία απλοποίηση της ε, ε, δαπάνης κονδυλίων μέσα από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι απαραίτητο ότι εάν φανεί ότι ότι είναι σαφής η ευθύνη των αρχηγών αντιπροσωπείων και των ε, υπαλλήλων της Επιτροπής Εξωτερικών Ενεργειών, αυτό δεν θα έδινε τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγξει την λειτουργία αυτών των κονδυλίων. Και υπενθυμίζω ότι το δικαίωμα του ελέγχου του προπολογισμού είναι από τα βασικά δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά. Χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιαστεβίτσιος. Πηγαίνουμε στο σημείο 5 τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την απαλλαγή από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα. Συγγνώμη. Α, μάλιστα. Είχε, πει και τα, είχε παρουσιάσει και τα δύο θέματα μαζί. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, τόσο το καλύτερο. Θέλει κάποιος άλλος να λάβει το λόγο. Όχι, κανείς. Θα ψηφίσουμε στις 9 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο για τις νομοδοτήσεις αυτές. Έχουμε τελειώσει τρία λεφτά νωρίτερα. Ο κύριος Βίγκαν δεν είναι ακόμα παρόν. Θα έρθει και ο εκπρόσωπος της Ουκρανίας. Μάλλον έχει έρθει ο πρέσβης της Ουκρανίας, τον οποίο ίσως μπορώ να δώσω το λόγο. Τα γεγονότα του Σαββάτου όπου έχασαν τη ζωή τους 13 άτομα στην Μαριούπολη είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός. Περιελάμβανε και ε, το ότι χρήση ρωσικού εξοπλισμού από τις αποσχιστικές δυνάμεις όπως ανέφερε και η ΟΑΣΕ την ε, Πέμπτη θα λάβει χώρα η, συνόδος, η συνάντηση των τεσσάρων Υπουργών Εξωτερικών και Έχω τονίσει τη σημασία της συμφωνίας για την απόσυρση των βαρέων όπλων ως μια προϋπόθεση για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η συνεννόηση για τα θέματα αυτά. Αυτό για πολλούς παρατηρητές πάντως στα γεγονότα του Σαββάτου δείχνει ότι οι αποσχιστικές δυνάμεις δεν είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις και έχουν την πρόθεση να εξαπολύσουν μια γενικότερη επίθεση σε όλη την περιοχή. Και φυσικά η Μαριούπολης είναι ένα κομβικό σημείο γιατί εξασφαλίζει και τον έλεγχο της Κρυμαίας. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη το, γεγονό, το γεγονός αυτό. Επομένως να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να παραμείνουν ρωσικά βαρέα όπλα στα χέρια των δυνάμεων αυτών που είναι αποσχεστικού χαρακτήρα. Έχουν μιλήσει οι αποσχεστικές αυτές δυνάμεις οι αντάρτες για μία ε, απελευθέρωση του ρωσικού πληθυσμού της Ουκρανίας και έχουν προβεί σε επιθετικές ενέργειες. Οι ενέργειες τους αυτές λοιπόν θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τις ε, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Εμείς ελπίζαμε ότι εφέτος θα μπορούσε να υπάρξει μια λύση στο πρόβλημα αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε το όλο πρόβλημα αυτό μετά από τα πρόσφατα γεγονότα. Έχουμε λοιπόν μια πολύ σοβαρή κρίση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην Ουκρανία. Το γεγονός ότι έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών καταδεικνύει τη σοβαρότητα αυτού του προβλήματος και η ανάλυση των Υπουργών έχει και ένα χαρακτήρα αρνητικό σε σχέση με ορισμένε επιλογές που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πώς μπορεί να συνεχίσει, πώς μπορούν να συνεχιστούν οι συνομιλίες στο πλαίσιο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί. Και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν τονίσει ότι με τη σταδιακή εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ μπορεί να εξομαλιστεί η κατάσταση, αλλά τώρα βλέπουμε ότι τα πράγματα μάλλον πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από την κατάσταση αυτή. Το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών έκανε σαφές ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστούν <clears throat> και να παραταθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αυτή ήταν η γενική άποψη. Αυτό <clears throat> δεν ίσως θα μπορούσε κανείς να το προβλέψει, αλλά παραμένει το ερώτημα αυτό και παραμένει το θέμα του αν θέλουμε όχι μόνο να παρατείνουμε τις ε, κυρώσεις, αλλά να τις ενισχύσουμε περαιτέρω. Θα μπορούσε λοιπόν το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών να ζητήσει από την Κομισιόν να διερευνήσει πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν περαιτέρω ε, κυρώσεις οι οποίες να καλύπτουν να τύχουν κυρίω τον οικονομικό τομέα. Καμία από αυτές τις εξελίξεις δεν μπορεί να θεωρηθεί θετική λοιπόν. Συμβαίνουν και πολλές ε, ενέργειες στην ε, Μολδαβία που ενδεχομένως μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι συνδέονται με αυτά τα γεγονότα. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει περαιτέρω αρνητικέ ε, ενέργειες στη Μολδαβία. Μέχρι πριν από μία εβδομάδα θεωρούσαμε ότι απλώς η περιχαράκωση και η συγκράτηση θα ήταν επαρκής. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει από τις αποσχιστικές δυνάμεις μια σαφής πολεμική διάθεση, μια επιθετική διάθεση. Υπάρχει παροχή βαρέως στρατιωτικού υλικού από την Ρωσία με το προσωπικό το οποίο εξυπηρετεί και ε, χειρίζεται αυτά τα βαρέα όπλα. Υπάρχει λοιπόν τακτικός ρωσικός στρατός στην Ουκρανία. Αυτή είναι η εντύπωση που εγώ έχω ε, διαπιστώσει και αυτό για μένα σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι πλέον. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε την ίδια αισιοδοξία που μπορεί να τρέχουμε στο παρελθόν. Δεν μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την ε, ε σχέση μας με την ε, Ρωσία <clears throat> και τις διαπραγματεύσεις μας για πολλά άλλα σημαντικά θέματα με τη Ρωσία παράλληλα με την ε, εξέλιξη αυτών των επιθετικών ενεργειών οι οποίες παραβιάσουν το διεθνές δίκαιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το οποίο πιστεύω πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και σε σχέση με αυτό δεν θα πρέπει να ε, ευνοήσουμε ένα κλίμα ψευδεστήσεων στη Μόσχα. Το ψήσιμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενεκρίθη στην Ολομέλεια ήδη είχε αναφερθεί και σε αυτήν την προβληματική και περιελάμβανε συγκεκριμένες αιτήσει από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να, να προτείνω να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Βίγκαν και μετά τον κύριο Έλιζεφ, τον πρέσβη της ε, Ουκρανίας, ο οποίος θα είναι σε λίγο και αυτός εδώ. Να ακούσουμε την ανάλυση του κύριου Βίγκαν και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση για το πρακτέον από εδώ και πέρα. Έχετε το λόγο, εξοχότατε. Το λόγο πρώτα στον ε, κύριο Παζευτή. Yeah, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Μπρόκ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Καταρχάς, ε, σας ευχαριστώ πολύ που έχετε συμπεριλάβει το θέμα της Ουκρανίας ε, στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα. Ο Ουκρανικός λαός ε, πλήττεται πάρα πολύ σοβαρά από την ε, ε, επεκτατική πολιτική της Ρωσίας. Οι ρωσικοί πύραυλοι εξακολουθούν να οδηγούν στο θάνατο ουκρανικές οικογένειες. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους και βρέθηκαν να ζετιανεύουν και να υποφέρουν. Τις τελευταίες ημέρες η Ουκρανία αντιμετώπισε κάποιες εξωφρενικές τρομοκρατικές πράξεις. Καταρχάς, βομβαρδισμός ενός λεωφορείου στην Όμπανχαν, πριν, μετά στο Ντόνετς και τώρα στη Μαριούπολη. Ε, μια πολυ, πυκνοκατοικημένη πόλη με περίπου 30 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά και πάνω από 100 τραυματίες. Ενώ 12.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή του βομβαρδισμού. Όλα αυτά συμβαίνουν ε, ενώπιον ε, άχαρων ρητορικών από ανθρώπων οι οποίοι δήλωσαν ε, το Σάββατο ότι μια επίθεση κατά της Μαριούπολης θα ήταν ο καλύτερος φόρος τιμής ε, για να ξεπληρώσουν το χρέο τους. Δεν υπήρχε καμία καταδίκη, κανείς δεν συλληπίθηκε ε, από πλευράς ρωσικής ηγεσία, απλώς κάποιες κοινικές δηλώσεις του Υπουργού Λαυρόφ, ο οποίος είπε ότι αν το Κίεβο είχε δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Πούτιν, αν θέλουμε το θεωρούμε ειρηνευτικό ε, το λέμε ειρηνευτικό σχέδιο, οι επιθέσεις στο Ντόνετ και στη Μαριούπολη δεν θα είχαν συμβεί. Το λεγόμενο σχέδιο που Πούτιν, απλώς για να σας το υπενθυμίσω, ήταν απλώς κατοχή ουκρανικών εδαφών και απώλεια κυριαρχίας. Επομένως το ερώτημα είναι αν η δήλωση του Λαυρόφ ε, είναι πραγματικά εκβιασμός. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αν η Ρωσία δεν είχε παραβεί την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας, δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή πόλεμο στην Ευρώπη. Αν η Ρωσία είχε αναλάβει τις ευθύνες της ε, για την τήρηση της των συμφωνιών του Μίνσκ, δεν θα υπήρχαν θάνατοι στην Ουκρανία. Αν η Ρωσία είχε σταματήσει την εισρωή ε, σε ε, ουκρανικά εδάφη ε, ρωσικών στρατευμάτων δεν θα υπήρχε ανάγκη και δεν θα υπήρχαν καθόλου βομβαρδισμοί κατοικημένων περιοχών από τρομοκράτες. Όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι η Ρωσία συμμετείχε στην προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων στις Ουκρανικές πόλεις, στην Οδυσσό, στη Χάρκιο, στο Μικολάιο και σε άλλες πόλεις η Ρωσία δεν παρέχει μόνο οπλισμό και στρατεύματα στα ουκρανικά εδάφη, αλλά βοηθά και σε τρομοκρατικές πράξεις. Το, κρίμ, ε, το έγκλημα της Μαριούπολης ε, κατά της ανθρωπότητας καθώς και πολλές άλλες τραγωδίες αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την τρομοκρατική φύση ε, των κατοίκων των, ρωσικών, των ρωσόφωνων περιοχών πρέπει να απαντήσουν στο δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία διέπραξαν τρομοκράτες το 2014 και το 2015, καθώς επίσης και την αναγνώριση ε, των ανθρώπων που δρούν εκεί ως τρομοκρατικές οργανώσεις. Πραγματικά πρόκειται για διεθνή τρομοκρατία. Όσο η Ρωσία συνεχίζει να υποσταλεί τους εγκληματίες και τρομοκράτες και τους δίνει τον πιο ε, προηγμένο βαρύ εξοπλισμό που ε, χρησιμοποιείται για επιθέσεις, σημαίνει ότι έχει ευθύνη για την κλιμάκωση της κατάστασης και για τα θύματα ε, που είναι απλοί πολίτες, επαναλαμβάνω, στον Ντενιέσκ, στη Μαριούπολη και σε πολλές άλλες ουκρανικές πόλεις και χωριά. Από σήμερα αυτά τα αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη ε, εχθροπραξίες στην περιοχή του Ντονιέσκ. Γι' αυτό ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει η Ρωσία τις επόμενες ώρες είναι τα εξής. Πρώτον, η Ρωσία θα πρέπει αμέσως να αναλάβει υπεύθυνε δράσεις ώστε να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Επίσης, η κυβέρνηση της Ρωσίας θα πρέπει προσωπικά και δημοσίως να καταδικάσει τους τρομοκράτες, διότι βομβάδισαν τη Μαριούπολη και να τους ζητήσουν να ακολουθήσουν τη λογική της ειρηνευτικής διαδικασίας βάσει των συμφωνίων του Μίσκ. Δεύτερον, η Ρωσία αναμένεται να ζητήσει από τους τρομοκράτες να σεβαστούν πλήρως τη συμφωνία. Τρίτον, θα πρέπει να συναντηθούν αμέσω με την τριμερή ομάδα επαφή για να συμφωνήσουν για τον τρόπο απόσυρση των στρατευμάτων βάσει του μνημονίου του Μίνσκ τη 15 η Σεπτεμβρίου του 2014. Τέταρτον, να διασφαλίσουν ότι οι τρομοκράτε ε, θα αποσύρουν τον βαρύ εξοπλισμό από τα σημεία επαφή. Τρίτον, να δώσουν ε, εντολή στι ε, ένοπλε δυνάμει τη Ρωσία να σταματήσουν τι επιθέσει του και να αποσύρουν τα στρατεύματά του από τα ουκρανικά εδάφη. Έκτον, να σταματήσει η ε, μεταφορά ως εξοπλισμού για προσωπική χρήση από τα σύνορα και να μην ε, αποτρέψουν τις Ουκρανικές αρχές να τις αφήσουν να αποκαταστήσουν την κυριαρχία τους στα σύνορα με τη Ρωσία και να αποκτήσουν πλήρη κυριαρχία βάσει ε, παρακολούθησης και από τον ΟΣΕ και επίσης θα πρέπει να απελευθερωθούν όλοι ε, οι κρατούμενοι και ε, όλα βάσει διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Οι τρομοκράτες που υποστηρίζουν από τη Ρωσία θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόσουν αμέσως τις συμφωνίες του ΜΕΣ και καλή την πίστη. Τι περιμένουμε εμείς κύριε Πρόεδρε από τη διεθνή κοινότητα. Πρώτον, να ενισχύσουν την πολιτική κυριώσεων και να τη διατηρήσουν για να μπορέσει να πιεστεί η Ρωσία να σταματήσει αυτές τις αποστερεοποιητικέ δράσεις. Επιπλέον μέτρα, όπως πολύ σωστά είπατε, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν χρηματικές κυρώσεις, ενεργειακές κυρώσεις, απαγόρευση για τη μεταφορά ε, οπλισμού, ε, να υπάρχουν απαγορεύσει θεωρήσεων διαβατηρίων ε, και να ζητήσουμε από τον πρόεδρο Πούτιν ε, να σταματήσει και να έχει για παράδειγμα και κάποιες κυρώσεις του τύπου απαγόρευση του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου της FIFA ε, στην επόμενη διετία. Επίσης να υπάρχουν ανθρωπιστική, οικονομική, ανθρωπιστική και φυσικά στρατιωτική συνδρομή. Και τρίτον, να υπάρχει συνεχής και επίμονη διπλωματική πίεση ώστε να υποχρεωθεί η Ρωσία να ξεκινήσει ένα αυθεντικό διάλογο. Παρά τις προκλήσεις η, Ρουκρία, η Ουκρανία δεσμεύεται, επαναλαμβάνω δεσμεύεται για μια ειρηνική λύση. Και αυτό είναι ο μόνο δρόμο προ την ειρήνη. Γι' αυτό ακριβώ και θεωρούμε ότι ε, η έκτακτη Σύνοδο του, Υπουργείου, του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, στο οποίο αναφερθήκατε και εσεί, κύριε Πρόεδρε, ε, η οποία θα δώσει κατευθύνσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Εξωτερική δράση και στα κράτη-μέλη να προετοιμάσουν μία δέσμη μέτρων και κυρώσεων κατά τη Ρωσία. Αυτό βάσει και του ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιανουαρίου του το 2015. Αυτό το οποίο σίγουρα δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει μια πιο ήπια πολιτική ε, και ε, ανοχή ενώπιον των Ουκρανικών αρχών. Αυτό θα διακυβάσει την εθνική κυριαρχία και την εδαφική κυριαρχία της χώρας μας και φυσικά θα ε, αυξήσει και την όρεξη του... Herzlichen Dank. Ich möchte Ευχαριστώ πολύ. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε. Η Ρωσία να δίνει την εντύπωση ότι δεν είναι εμπλεκόμενη στη σύγκρουση. Είναι τμήμα της σύγκρουσης η Ρωσία. Είναι μία από τις δυνάμεις οι οποίες εμπλέκονται στις εχθροπραξίες. Θα πρέπει λοιπόν να ξεχάσουμε τις παλιές μεθόδους της ΚΑΓΕΜΠΕ της ε, απόκρυψης και της ε, δημιουργίας εντυπώσεων οι οποίε δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Κύριε Βίγκαν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και πρόεδρε. Αν μπορώ να έρθω στο τελευταίο σα σχόλιο. Θα ήθελα να σταθώ στην σαφή δήλωση η οποία έγινε από την ύπατη εκπρόσωπο μετά από τα γεγονότα της Μαριούπολης το Σάββατο η κυρία Μπογκερίνη τόνισε τη σημαντική επιρροή που ασκεί η Ρωσία στους ηγέτες των αποσχιστών και ζήτησε από τη Ρωσία να σταματήσει οποιαδήποτε στρατιωτική, πολιτική ή οικονομική υποστήριξη για τους ηγέτες των αποσχιστικών δυνάμεων. Αναφέρθηκε επίσης η τραγική απόλυξη του βομβαρδισμού της Μαριούπολης που στήξε 13 ζωές αμάχων και τόνισε ότι μια τέτοια ενέργεια δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε περαιτέρω επιβάρυνση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Όπως είπε ο πρεσβευτής κ. Σελισέβες, δεν μπορεί να υπάρξει μια ειρηνική επίλυση αυτή τη στιγμή και η κυρία Μογκερίνη, η υπατή συνεκάλεσε ένα έκτακτο συμβούλιο υπουργών εξωτερικών για να επιληθεί του θέματος αυτού όπως ελέγχθη, έχει συνεχιστεί μια κατάσταση που οδηγεί σε άμαχα θύματα. Είναι ένα τραγικό ε, γεγονός σε μια χρονική εποχή που πρόκειται να υπάρξει αποκλιμάκωση της ε, σύγκρουσης. Υπάρχει λοιπόν εντατικοποίηση των στρατιωτικών δράσεων και αυτό συνοδεύεται από περαιτέρω δηλώσεις επιθετικού χαρακτήρα από τις αποσχεστικές δυνάμεις. Θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση με τον καταλληλότερο τρόπο στις ε, προκλήσεις αυτές από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση θα πρέπει να επιληφθεί και να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου. Οι Ουκρανικές αρχές έχουν τονίσει ότι οι αποσχεστικές δυνάμεις έχουν την υποστήριξη ρωσικών δυνάμεων και υπάρχουν περίπου 2.000 στρατιώτες που έχουν έρθει ε, από την Ρωσία στην περιοχή του Ντόνμπας με ε, εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Είχαμε και άλλα ε, γεγονότα στο Χάρκοβο, στο Μπομπλάς και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Υπήρξε εκτοχιασμός ενός φορτηγού εμπορικού τρένου, καταστράφηκε μία σιδηροδρομική γέφυρα. Όλα αυτά είναι σημάδια κλιμάκωσης και όχι αποκλιμάκωσης. Ο πρόεδρος Ποροσέγκο έχει κηρύξει μερική επιστράτευση που θα πρέπει να επιχειρωθεί από το Κοινοβούλιο και προβλέπεται να υπάρξει ε, κινητοποίηση μέχρι 100.000 εφέδρων. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 900.000 εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα στην ε, Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης ενισχύσει σημαντικά την ανθρωπιστική της βοήθεια προς την Ουκρανία, <clears throat> η οποία θα γίνει ιδιαίτερα ε, ορατή με την ε, επίσκεψη του Επιτρόπου Σιλιανίδη στο Νίπιο Πετρόφσκ για να τονιστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με μεταφορά και παράδοση φορτίων ανθρωπιστικής βοήθειας και σε περιοχές που δεν βρισκόνται υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Αυτό θα περιλαμβάνει και τη Μαριούπολη. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και είναι πάρα πολύ σημαντική και η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει κουπόνια τα οποία αντικαθιστούν το ρευστό χρήμα για να βοηθήσει τους πιο ενδέει στην περιοχή αυτή. Συνεχίζονται λοιπόν οι ενέργειες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρόφωνο παρακαλώ, Παρά τις ε, θετικές δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν στο Βερολίνο μετά από την συνάντηση 12 Νοεμβρίου, δυστυχώς η κατάσταση επιτοπίως δεν έχει εξελιχθεί με τον προσδοκόμενο τρόπο. Συνεχίζονται λοιπόν οι προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο για την απόσυρση βαρέων όπλων από την, από την γραμμή αντιπαράθεσης μαζί με μια κατάπαυση του πυρός. Δυστυχώς η ρητορική σε πολιτικό επίπεδο δεν οδήγησε σε συγκεκριμένες συνέπειες από αυτούς οι οποίοι υποστηριζόνται από τις ρωσικές δυνάμεις. Η ύπατη εκπρόσωπος μίλησε αυτή τη βδομάδα με τον πρόεδρο Ποροσέγκο της Ουκρανίας και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας τον Σεργέη Λαύροφ μεταδίδοντας αυτό το μήνυμα το οποίο προέρχεται από τη δήλωσή της 24ης Ιανουαρίου. Σήμερα συνεδριάζει το μόνιμο Συμβούλιο της ΟΑΣΕ. Θα έχουμε μια ειδική συνεδρίαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και έχουν ξεκινήσει και συζητήσεις στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με την ενδεχόμενη άρση των δικαιωμάτων ψηφοφορίας της ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας, αν θα πρέπει μάλλον να επανέλθουν αυτά τα δικαιώματα ή να παραμείνουν εκκρεμωτήτη. Όλα αυτά λοιπόν είναι απόρριες αυτής της πάρα πολύ απότομης επιδείνωσης κατάστασης. Επίσης κύριε Πρόεδρε, εάν μου επιτρέπετε θέλω να επιστήσω την προσοχή των μελών της Επιτροπής στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Γιατί όσο γίνονται όλα αυτά τα γεγονότα, έχουμε μια νέα κυβέρνηση στην Ουκρανία, η οποία είναι προσιλωμένη στι μεταρρυθμίσει που αναμένει η Ευρώπη και η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει την υποστήριξή της, η οποία εξαρτάται από τις μεταρρυθμίσεις. Ο νόμος περί προϋπολογισμού του 2015 ενεκρίθη το Δεκέμβριο και αντανακλά τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης. Περιλαμβάνει και στοιχεία αποκέντρωσης του φορολογικού συστήματος που έχουν μεγάλη σημασία. Προβλέπεται αναθεώρηση του πακέτου του προϋπολογισμού μέχρι 15 Φεβρουαρίου για να ληφθούν υπόψη νέες δεσμεύσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την διεθνή κοινότητα που θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτές τις προσπάθειες και ξέρετε ότι το Συμβούλιο συζητά τώρα για ένα νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής αρρωγής ε, για την Ουκρανία και το Ευρωπαϊκό Τμήμα αυτής της ενέργειας θα έλθει και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει μεταρρύθμιση του εκλογικού δικαίου που δεν έχει ακόμα καταλήξει σε μια πλήρη ενοποίηση της νομοθεσίας για τις εκλογές, αλλά η νομοθεσία για τις τοπικές εκλογές θα είναι έτοιμη πολύ σύντομα, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό για τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Υπήρξαν τροπολογίες οι οποίες έχουν ε, υποβληθεί από τον κύριο Ποροσέγκο μετά την εκλογή του, αλλά δεν έχουν ακόμα ψηφιστεί. Υπάρχει η αξιολόγηση Επιτροπής Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και ελπίζουμε ότι αυτή η αξιολόγηση θα κατευθύνει περαιτέρω προσπάθειε μεταρρυθμίσεω. Από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων να δημιουργηθεί πολύ σύντομα, να είναι μια περιεκτική ε, διαδικασία η οποία θα αντιμετωπίσει και όλα τα θέματα αποκέντρωση, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και ένα περιεκτικό εθνικό διάλογο που είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του μηνύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία που ζητά να υπήρξουν να υπάρξουν και εσωτερικές ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία αναδύθηκαν στη διάρκεια της κρίσης. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς υπήρξαν πολλά μέτρα τα οποία λύθησαν με μια δέσμη μέτρων κατά της διαφθοράς που ενεκρίθη από το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας και που συμπεριλαμβάνουν ένα νέο νόμο κατά της ε, ε, ε, δημιουργία επιτροπής καταπολέμησης της ε, διαφθοράς και είναι ο, πρόεδρος, ο επικεφαλής ΟΛΑΦ πρόεδρος της Επιτροπής που έχει σαν στόχο να δημιουργήσει αυτή τη νέα Επιτροπή κατά της διαφθοράς. Θέλω λοιπόν να τονίσω και δύο ακόμα δύο νομοθετήματα για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσίας που συζητήθηκαν στην, στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο στις 13 ε, ε, Ιανουαρίου. Η Βέρχο Βαράντα έχει δημιουργήσει μια επιτροπή η οποία εξετάζει τις δύο αυτές προτάσεις του Προέδρου της Ουκρανίας και μιας ομάδας κοινοβουλευτικών και θέλουμε να ζητήσουμε από τους Ουκρανούς ομολόγους μας να εξασφαλίσουν ότι οι κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και αυτής της Επιτροπής θα πρέπει να ληφθούν ε, υπόψη. Επίσης, για τις τηλεοπτικές εκπομπές, στις 13 Ιανουαρίου <clears throat> το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας πέρασε νομοθεσία για τις δημόσιες εκπομπές και ζητήθηκε επίση από τον πρόεδρο τη Βουλή να λάβει περαιτέρω τροπολογίε εν ώψη που να προέρχονται από τον, πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο τη επιτροπή για την Ελευθερία των Μέσων ενημέρωση. Έχουμε κάποιε ανησυχίε στον χώρο αυτό. Θα θέλαμε να έχουμε να έχουμε μια ανεξάρτητη ραδιοτηλεοπτική επιτροπή η οποία να έχει ανεξαρτησία στην Ουκρανία. Θέλω επίση να σα υπενθυμίσω ότι όλο αυτό είναι η απαρχή μια μεγαλύτερη διαδικασίας μεταρρύθμισης όπως αναφέρεται στη Συμφωνία για το Κυβερνητικό Συνασπισμό και στην Εθνική Σύλληψη για τη Μεταρρύθμιση που σύντομα θα ε, υλοποιηθεί, θα έχει διατυπωθεί καλύτερα και θα είναι το αντικείμενο μιας διεθνούς συνδιάσκεψης. Η υποστήριξη λοιπόν σε όλες αυτές τις ενέργειες γίνεται από την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μια αποστολή ΚΕΠΑ Έχοντας πει όλα αυτά, θέλω να κλείσω. Αν έχετε και ερωτήματα, είμαι έτοιμος να δώσω απάντηση για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέω ο πρόεδρος, χωρίς το μικροφωνό του βέβαια. Είναι 14 συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο. Θέλω να σας παρακαλέσω λοιπόν να είσαστε σύντομοι και κλείνω τον κατάλογο αγορτών. Σας παρακαλώ να περιοριστείτε στο ένα λεπτό. Ο κύριος Πλένκοβιτς είναι ο πρώτος ομιλητής. Ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ουκρανία. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε Μπρόκ και σας ευχαριστώ. Εγώ σας ε, συγχαίρω για το γεγονός ότι συγκαλέσατε τη σημερινή συνεδρίαση με θέμα την Ουκρανία. Ε, την περασμένη εβδομάδα μιλούσαμε με τον κύριο Γελισέγεφ ε, ε, σχετικά με την επιδεινούμενη κατάσταση. Καταδικάσαμε την τρομοκρατική επίθεση στη Μαριούπολη όπου υπήρξαν τόσα θύματα άμαχου πληθυσμού. Πραγματικά εκφράζονται τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και στην Ουκρανία. Ε, είναι αυτή η ευκαιρία να στείλουμε ένα στεναρό μήνυμα στην Ρωσία και να ε, εντείνουμε τα μέτρα πίεσης γιατί υπάρχει σαφή σύνδεση ε, με το μεταξύ τρομοκρατικών επιθέσεων και των αποσχιστικών που στηρίζονται από το Κρεμλίνο από τη Ρωσία. Πιστεύω ότι την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε μια συζήτηση για την προετοιμασία μιας πρώτης επιτροπής σύνδεσης που θα γίνει εδώ στο Βρυξέλλες και προσβλέπω στη συμβολή όλων των συναδέλφων για αυτή τη συζήτηση στην... για την Ουκρανία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω, δεδομένου ότι η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά, νομίζω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να επιβάλλουμε μια διαπραγματευτική λύση. Γιατί κάθε φορά που διαφαίνεται μια διπλωματική λύση στον ορίζοντα, πάντα υπάρχει κάποιο, και κυρίω ο Πούτιν πρώτο και καλύτερο, που προσπαθεί ε, να υψώσει κι άλλο τον πύχη. Ε, και αυτέ τι ε, μέρε έκανε επίδειξη αυτή τη τακτική. Πιστεύω πω είναι σημαντικό από τη μια πλευρά βεβαίω, δεν θεωρούμε αποδεκτό όσα έγιναν για την Κρυμαία και κυρίως τι συνεχιζόμενες παρεμβάσει στην ανατολικό τμήμα τη χώρα από πλευρά τη Μόσχα. Ωστόσο δεν θα πρέπει και να ξεχνάμε τα σφάλματα που έχουν ε, γίνει σε σχέση με κάποιε προσδοκίε που καθορίστηκαν και όσον αφορά το θέμα της ευρωπαϊκής ένταξης, της εισόδου στο ΝΑΤΟ και τι καθυστερήσεις δηλαδή και στι μεταρρυθμίσεις. Η γνώμη μου λοιπόν είναι σχετικά ότι πρέπει να εντοπίσουμε τα μέρη τα οποία μπορούν να επιβάλλουν ε, μια λύση ε, και είναι η ΕΠΑ ε, και η Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να βρει μια εσωτερική συνοχή από μια πλευρά θα πρέπει να βάλουμε στην άκρη και τις επιθυμίες εκδίκησης και, και τη δηλία μας που που έχουμε δείξει μέχρι στιγμή. Θα είναι μια πρώτη μεγάλη ε, δοκιμασία για να μπορέσουμε να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Χρειάζεται θάρρος και αποφασιστικότητα. Πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Ο κύριος Στάνοκ, σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω καταρχήν εξ ονόματος της ομάδας μου ε, τα συλληπιτήριά μας ε, στις οικογένειες των θυμάτων και στην Ουκρανία γενικότερα ε, για τα θύματα, όπως είπα, τη τελευταία τρομοκρατική επίθεσης. Πρόκειται για μια ηθελημένη επίθεση σε κατοικημένες περιοχές μέσω πυράβλων και βομβαρδισμών. Πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση που στόχο έχει να τρομάξει, να τρομοκρατήσει τον, ε, τους πολίτες σε 30 θάνατοι, παιδιά, γυναίκες, ε, εκατοντάδες θύματα και τραυματίε. Στην ουσία σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου κάτι τέτοιο θεωρείται έγκλημα πολέμου. Και γι' αυτό και καλωσορίζω την παραπομπή του Αρκείου στο Δικαστήριο Ποινικού το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ελπίζω ότι θα διερευνηθεί πλήρως ε, αυτή η κατάσταση και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτές τις φρικαλαιότητες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, ιδιαίτερα εκείνοι ε, που έχουν δράσει σε αυτές τις περιοχές. Ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει το αμερικανικό παράδειγμα, να κλιμακώσει και να εντείνει το καθεστώς των κυρώσεων απέναντι στο καθεστώς της Μόσχας, ε, κυρίως όσον αφορά τα εμβάσματα SWIFT, δηλαδή να μην μπορούν πλέον ε, οι Ρώσοι να δουλέψουν με τις δικές μας επιχειρήσεις ε, και βέβαια θα καλέσω τα μέλη του ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν αυτό που κάνει και η Ρωσία, δηλαδή να δίνουν στους Ουκρανούς ένα, ένα κυρίαρχο κράτος με τα στρατιωτικά μέσα να υπερασπιστεί τον αυτό του απέναντι στη Ρωσία. Κάποια τάγκ όπως το Άμπραμ, το λέω παρτού, δεν θα έκαναν, δεν θα ήταν άσχημα. Πάντως πραγματικά η καρδιά μου θλίβεται για τους ε, αθώους πολίτες που έπεσαν ε, σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να αναφερθούμε στα γεγονότα. Η Κρυμαία είναι ακόμα κατεχόμενη υπάρχει ακόμα ρωσική παρέμβαση στην Ανατολική Ουκρανία και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα επεισόδια στη Μαριούπολη και στην ευρύτερη περιοχή που θα πρέπει να έχουν συνέπειες και νομίζω ότι η ύπατη εκπρόσωπος θα πρέπει να προτείνει στους Υπουργούς Εξωτερικών μια δέσμη κυρώσεων ε, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένε κυρώσεις, γιατί αυτό είναι απαράδεκτο. Η Ρωσία είναι επιθετική, οι συμφωνίες του Μουίνσκ έχουν μπει στο ράφι, λες και είναι ένα παλιόχαρτο και επομένως θα πρέπει να δράσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είπα, ότι εκπρόσωπος να ε, κάνει προτάσεις και οι υπουργοί να συμφωνήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο θάνατος ε, αθών πολιτών ε, σε ε, στρατιωτική σύγκρουση είναι λόγος για να αλλάξει το θεματολόγιό μας και μάλιστα να καταδικάσουμε καταρχάς αυτές τις τηλεφωνίες και οι ένοχοι να πληρώσουν, αλλά για τα πάντα. Διότι πρέπει να πω ότι συγκεκριμένη αλλαγή δεν είμαι βέβαιος ότι έχει γίνει έτσι. Υπήρξε δελτίο τύπου του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος επεσήμανε ε, ότι θα πρέπει, ε, ε ότι ε, την ε, Ρωσία για την ε, κατάσταση αυτή. Ε, ο καθένας έχει τις προτεραιότητες. Έχει γίνει ένα πανδεμόνιο κατά της Ρωσίας η Επιτροπή μας στη διάρκεια αυτής της θητείας είναι αδύνατο να κάνουμε μια λογική ανάλυση αυτή τη στιγμή. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε μια οβίδα η οποία έχει ε, παγιδεύσει 500 ανθρακορίχους ε, σε ένα ανθρακοριχείο στον Τόνεξ αυτή τη στιγμή. Και επομένως ε, θα πρέπει να τα τονίσουμε αυτά τα πράγματα. Και λυπάμαι πολύ για την κατάσταση, όχι μόνο για το τι σημαίνει για τη Ρωσία, αλλά γιατί και εμείς πραγματικά προσπαθούμε να διευκολύνουμε αυτούς που μας θέλουν να μας απομακρύνουν από τους γείτονές μας και δεν προσπαθούμε να βρούμε μια ειρηνική λύση ως ένδειξη καλής γειτονίας. κύριος Κύριε Πρόεδρε, Μέζεριτ, συγγνώμη. Καταρχάς, ε, να συμφωνήσουμε με τα όσα είπε ο εκπρόσωπος της υπάτης εκπροσώπου και φυσικά να συλληπιθούμε και εμείς ε, στην οικογένεια των θυμάτων, κυρίως στη Μαριούπολη, αλλά γενικότερα στην Ανατολική Ουκρανία. Επίσης, καλωσορίζουμε το γεγονός ότι θα υπάρξει ένα έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και είμαστε βέβαιοι, απόλυτα βέβαιοι, ότι τώρα περισσότερο από ποντά χρειάζεται να μιλούμε με μία φωνή από πλευράς Ευρώπης. Δάλος, η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να παίζει αυτό το παιχνιδάκι για όσο χρόνο επιθυμεί. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν με ποιον συνομιλούν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πλευρά Ευρώπης. Αυτό το οποίο προκύπτει λοιπόν από εδώ, σαφέστατα, είναι ότι θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα κάνει στο εγγύς μέλλον κανένα κράτος μέλος ε, άμεσες συζητήσει συζητήσεις σε υψηλό επίπεδο με τη Ρωσία πριν υπάρξει οποιαδήποτε αποκλιμάκωση. Ακόμα και αν είναι ε, μεγάλη ή μικρή χώρα, είτε είναι η δική μου χώρα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως θα ήθελα να επαναλάβω, ε, συλληπούμαστε όλα τα θύματα και ε, αυτά είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και σίγουρα πρέπει να διαρευνηθούν και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σάιρους Βόλσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτον. Αυτό το οποίο έγινε στη Μαριούπολη δεν είναι κάτι το εκπληκτικό, είναι κάτι το οποίο ήταν προβλέψιμο. <clears throat> Δεύτερον, βρίσκω παράξενες διατυπώσεις σε αυτά που είπε η κυρία Μογγερίνη, ο κύριος Σούλτς και ο κύριος Ελισιάφεφ. Είναι ουσιαστικά αφελές και αντιπαραγωγικό το να ζητάμε από τη Ρωσία να ασκήσει πίεση στους ε, στις δυνάμεις. Έτσι ενισχύουμε τη ρωσική προπαγάνδα. Το μόνο το οποίο έχει νόημα είναι το μήνυμά μας να μην απλώς καταδικαστικό αλλά να οδηγήσει σε δράση χωρίς δράση θα είναι πραγματικά αντιπαραγωγικό να έχουμε οποιοδήποτε νέο κείμενο. Λυπάμαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απαλύνει το ψήφισμά του σε σχέση με το ψήφισμα του Σεπτεμβρίου 2014 μη αναφερόμενο στο SWIFT και λυπάμαι για το έγγραφο της 19ης Ιανουαρίου από την ύπατη εκπρόσωπο που ζητά μια αποκλιμάκωση της έντασης, όλα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι μια <clears throat> αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε περισσότερες κυρώσεις, ένα σύστημα ε, συνομιλιών Γενέβης και όχι τύπου Νορμανδίας. Χρειαζόμαστε παραδόσεις όπλων από το ΝΑΤΟ ή από κράτη-μέλη για να δώσουμε στην Ουκρανία τη δυνατότητα να ε, ε, μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αλλιώς η Ρωσία θα συνεχίσει την ε, επέλασή της μέχρι την υπερδυστερία και τέλος οι δημοκρατίες του Ντόνεσκ και του Λουχάνσκ πρέπει να θεωρηθούν τρομοκρατικές οργανώσεις. I'd like just to um, join my voice to those who are not by... Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι δεν με εκπλήσουν οι ρωσικές πράξεις και η υποκρισία όχι μόνο της Ρωσίας αλλά ακόμα και η δική μας. Ε. Από το δικό μας το στρατόπεδο που είναι στο μισθολόγιο της Gazprom ή οποιαδήποτε άλλη και αρνούνται να δουν την πραγματικότητα. Συμφωνώ λοιπόν με αυτούς που είπαν ότι γίγαινε η ώρα να δράσουμε και όχι απλώς να μιλούμε. Και δράση σημαίνει κυρώσεις, σημαίνει να δηλωθεί σαφέστατα ποιος είναι αυτός ο οποίος επιτίθεται. Και να δηλώσουμε ότι δεν είναι μια δράση η οποία ξεκινά εκ των έσω ε, και έχουμε αυτές τις ε, δολοφονικές επιθέσεις. Υπάρχει σαφέστατη ρωσική παρέμβαση και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να υποκρινόμαστε ότι δεν είναι τα πράγματα ως έχουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ε, κυρία Φωτίγκα, ευχαριστώ κύριε Πρέσβη για τα όσα μας είπατε σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας. Συμφωνώ απολύτως με πολλά από τα οποία ακούστηκαν σήμερα. Ο κύριος Στάνοκ, ο κύριος Άριος Βόλσκι, ο κύριος Βαμβάλεν, η κυρία Ναγκόμεζ, Νομίζω ότι είναι προφανές ότι πρέπει να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Και θα πρέπει πραγματικά να επανεξετάσουμε την ε, πολιτική μας ε, του καρότου και του μαστιγίου. Μάλλον παρά τα καρότα πολλά ή πολλές υποσχέσεις για καρότα. Επομένως θα πρέπει και εμείς ε, να σκεφτούμε τι κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να έχουμε ένα επίπεδο κυρώσεων αντίστοιχο των μέτρων της Ρωσίας. Οι κυρώσει θα πρέπει να είναι ε, πιο αυστηρές και θεωρώ ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να γίνει αυτό. Έχουμε πει ότι όταν να αποφασίσει η Ρωσία να προχωρήσει τότε θα πρέπει και εμείς να αυξήσουμε τις κυρώσεις μας και νομίζω ότι η Ρωσία προχώρησε και μάλιστα πολύ. Επομένως και εμείς θα πρέπει να τηρήσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε δεν θα πρέπει να ξεχνούμε για παράδειγμα την Κρυμαία. Πρόκειται για κατεχόμενη περιοχή και υπάρχει ένας υβριδικός πόλεμος σε μία γείτονα χώρα. Επομένως θα πρέπει και εμείς να κάνουμε αυτά τα οποία δηλώνουμε και να υπάρχει και υποστήριξη. Ευχαριστώ. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε όλοι μάρτυρες όλο και πιο μεγάλης επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αυτό που έγινε στη Μαριούπολη, δείχνει δυστυχώς ότι η Ρωσία δεν έχει καμία διάθεση να σταματήσει αυτές τις ενέργειες. Πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες ε, κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, γιατί κάθε φορά βρίσκει τρόπους να τις ε, παρακάμψει. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία απειλεί, εάν δεν άρουμε τις ε, να καταλάβει το Κίεβο, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε ένα Έχουμε μια υποχρέωση πολιτική και ηθική να περάσουμε από τις κυρώσεις σε, μποϊκότ, σε μποϊκοτάρισμα των ρωσικών προϊόντων και των αθλητικών εκδηλώσεων. Εμείς δυστυχώς δεχτήκαμε να είμαστε τμήμα των Ολυμπιακών του Σότσι και βλέπουμε ότι μετά από το 2018 θα υπάρξουν πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα οποία εμπλέκουν την Ρωσία. Αν είμαστε σοβαροί ας κάνουμε περισσότερες κυρώσεις. Περισσότερα για περισσότερα αυτό πρέπει να είναι η αρχή μας. Και να ελευθερωθεί η Νάντια Σέτσενκοφ η οποία κρατάται παράνομα από τους επιτιθέμενους Ρώσους και θα πρέπει να ελευθερωθεί γιατί είναι η ηρωίδα της Ουκρανίας. Um, um, Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Από την εποχή του, της συμφωνίας του Μίνσκ υπάρχουν συνεχείς ψευδεστήσεις σε σχέση με την πολιτική που ακολουθεί η Ρωσία. Παράξενες ιδέες χώρες οι οποίες βρίσκονται σε διμερείς συζητήσεις με τη Ρωσία και αγνοούν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας με, με χήμερες και ψευδεστήσεις να θεωρούμε ότι μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε με τη Ρωσία. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι αδύνατο. Πρέπει να προχωρήσουμε να μην άρουμε τις κυρώσεις, θα πρέπει να τις ενισχύσουμε οι υποστηρικτές του κυρίου Πούτιν πρέπει να τεθούν σε μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το σύστημα SWIFT. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Ρωσία θα απομονωθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης. πρέπει να υποστηρίξουμε την, ε, Ουκρανία με τεχνογνωσία και με εξοπλισμό. Οι λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες στο Λουγκάνσκ και στο Ντόνιασκ θα πρέπει να αναφερθούν ως τρομοκρατικές οργανώσεις. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει την επίθεση μιας πιο ισχυρής στρατιωτικής δύναμης που δίνει βαριά όπλα και πυρομαχικά στους, στις αποσχετικές δυνάμεις εκεί. Πρέπει εμείς να υποστηρίξουμε την Ουκρανία που είναι θύμα επιθέσεως. Κύριε Μπρόκ, είπατε και εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι η Ρωσία είναι τμήμα της σύραξη. Είναι πολύ περισσότερο. Πρόκειται για μια σύραξη η οποία δεν μπορούμε να πούμε ούτε ρωσική ούτε επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Είναι μια σύγκρουση στην οποία παρεμβαίνουν και είναι και ένα απόσπαστο τμήμα της Ουκρανία. Τώρα, το γεγονός ότι οι Ουκρανοί, οι οποίοι παρεμβαίνουν ε, από πλευράς επιμελητίας και επιχειρησιακής, κατευθύνονται από τη Ρωσία. Γι' αυτό εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά το να λέμε ότι υπάρχει εξωτερική επίθεση κατά μιας χώρας, σημαίνει ότι λησμονούμε ότι υπάρχουν εσωτερικοί παράγοντες. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας επίθεσης. Αυτό είναι σαφές για μένα. Επίσης είναι σαφές ότι υπάρχει δάκτυλος της Ρωσίας. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για στρατηγικές αναλύσεις για το ποιος είναι υπεύθυνο ε, και, ε, και να ξεχνάμε ότι πρέπει εμείς να αναλάβουμε μέτρα. Εγώ θεωρώ ότι η Ρωσία είναι τμήμα της σύγκρουση και για μένα αυτή είναι μια περίπτωση ε, στην οποία ακούμε μόνο τη μία πλευρά. Δεν θέλω να τι θέσω επίση όρει, διότι είναι σαφέ ότι η Ουκρανία είναι το θύμα και η Ρωσία είναι επιτιθέμενο. Αλλά η Ρωσία υπάρχει, είναι μια υπερδύναμη και εδώ κανεί δεν ακούει τη Ρωσία. Εγώ δεν ε, ε, δεν έχω ακούσει ποτέ η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να προσκάλεσε κάποιον και να ακούσουμε εδώ τη Ρωσία για να δούμε τι έχει να μα πει. Όχι για να συμφωνήσουμε με τη Ρωσία, αλλά για να δούμε τι έχει να μα πει. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πριν από χρόνια ε, μίλησα με έναν υπεύθυνο ε, σχέσεων επικοινωνίας ε, του Ισραηλινού στρατού, του στρατηγού Φρέμες Νεφ. Μου είπε, κοιτάξτε, η ειρήνη γίνεται με τους εχθρούς και πρέπει να τους ακούσουμε και αυτούς. Και σε αυτή την περίπτωση αναφερόταν στους Παλαιστινίους που θεωρούνταν τρομοκράτες. Ας ακούσουμε λοιπόν, διότι δεν μπορούμε να έχουμε εξωτερική πολιτική απλώς ε, συζητώντας μεταξύ μας κατά συνέπεια το να υπάρχουν καταδίκες και να υπάρχουν απλώς ε, ε, ισχυρισμοί ε, το μόνο που μας μένει για να είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας είναι να κηρύξουμε πόλεμο κατά της Ρωσίας και νομίζω ότι αυτό είναι δυσανάλογο. Αυτό δεν σημαίνει και με αυτό ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε ότι είμαι με τη Ρωσία, ίσα ίσα που είμαι κατάφορα αντίθετος, αλλά είμαι αντίθετος επίσης και στο να ακούμε απλώς μόνο τη μία πλευρά. Oui, ça Usama. Monsieur le Président, euh, je pense... Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι δικαίως δικαίως ε, ε, εμείς ε, ε, ασχολούμαστε με την υπόθεση της Μαριόπολης ε, ε, αλλά θα ήμασταν πιο ειλικρινεί αν ε, πριν 10 μέρες είχαμε την ίδια στάση με το ε, μαζικό βομβαρδισμό του Τόναξ. Δηλαδή δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε διαφορετικά μέτρα και σταθμά και να έχουμε μια επίθεση δίκαιη και θεμετή που προσανατολίζεται μόνο προς μια κατεύθυνση, αλλά δεν έχει καλούς νεκρούς και κακούς νεκρούς από την άλλη. Έπειτα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και το γνωρίζετε. Έχω ένα παράδειγμα και ε, απόδειγμα ε, απόδειξη μάλλον ότι υπήρξαν χειραγώγηση. Ο Ιζιμπέκοβιτς ενώπιον του κυρίου Κουσνέρ δέχεται ότι χειραγώγησε τα γεγονότα. Ε, ε, έχουμε τα γεγονότα στη Μισοάρα και αλλού και το, ξέρω στην ιστορία εκατοντάδες παραδείγματα χειραγώγησης. Ας μην δρούμε λοιπόν μόνο στα, στα γεγονότα χωρίς να ε, βλέπουμε ολόκληρη την εικόνα και να χρησιμοποιούμε την ευθεία μας. Το να, το να τους βγάλουμε από το SWIFT πρόκειται για κίνηση πολέμου. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που έχει την πυρηνική ναι, ε, βόμβα. Μα αυτό σημαίνει όμως ε, τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που θα είναι πυρηνικός. Δεν συνειδητοποιείται τι κάνετε γιατί δεν θέλετε δεν θέλετε να έχετε την ε, πλήρη εικόνα μιας ε, κατάστασης. Δεν, ε, δεν είναι όλα άσπρο μαύρο, όλα από εδώ και σωστά και όλα από εκεί λάθος. Δεν ετοιμάζουμε έτσι την ειρήνη. Mr. Gala. Thank you very much. I Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να καλέσουμε τον πρόεδρο Τσίσοφ την ιδέα που είχε ο συνάδελφος ε, αν και ξέρω τι θα μας πει, αλλά υπάρχει κάποιος σε αυτή την αίθουσα που να πιστεύει ναι, συγγνώμη. Υπάρχει κανείς σε αυτή την αίθουσα που να πιστεύει ότι ένα τάγκ ή ένας και μόνος στρατιώτης θα διασχίσει τα ουκρανικά σύνορα χωρίς την έγκριση του Ρώσου Προέδρου. Ας πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αυτός χρειάζεται τη σύγκρουση και τα εδαφικά παιχνίδια για να αιτιολογήσει το κοινωνικό κόστος του πολέμου του στην χώρα του. Δηλαδή η καταβήθηση του προγράμματος συνταξιδότησης για να χρηματοδοτήσει την Κρυμαία 400 ε, και ένα σωρό νεκροί Ρώσοι στρατιώτε σύμφωνα με την Επιτροπή των Ρωσίδων Μητέρων. Την Πέμπτη λοιπόν θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένε προτάσει από την κυρία Μογκερίνη για επιπλέον κυρώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych Σα ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι πριν δύο μέρες, <coughs> προχτέ δηλαδή, ήταν η 20 επέτειος του θανάτου του Winston Churchill και θα ήθελα να σας θυμίσω τι έλεγε. Ότι ό,τι ποια συνθήκη υπογράφει κανείς με τη Ρωσία κοστίζει απλά και μόνο το χαρτί επί του οποίου τυπώθηκε. Και εξακολουθεί να ισχύει αυτό και σήμερα, κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε, διότι χωρίς διαπραγμάτευση δεν μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος οποιασδήποτε σύγκρουσης. Όμως όσον αφορά τις κυρώσεις, ναι, πρέπει να γίνουν και άλλες κυρώσεις, να γίνουν και άλλα βήματα. Στην τελευταία σύνοδο του Στρασβούργου ε, γκρίναμε το ψήφισμα για την Ουκρανία που λέει στο σημείο 14 ότι τίποτε δεν θα σταματά τα ε, κράτη-μέλη της Ένωσης από το να, να δίνουν μάλλον όπλα ε, και να προμηθεύουν την Ουκρανία με όπλα και σε δικό εξοπλισμό. Και ήθελα να κάνω έκκληση στα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα στη χώρα μου, την Τσεχία και τον Πρωθυπουργό της Τσεχίας, διότι η Τσεχία πρόσφατη έδωσε όπλα τους ε, πέσμεργάς του Κουρδιστάν, 250 τόνοι πυρομαχικών και ρωτώ τον Πρωθυπουργό της χώρας μου, ποια είναι η διαφορά της καταπολέμησης ε, του τρομοκρατίας των Πέσμεργάς και της Ουκρανίας. Ευχαριστώ. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je serai très, très court, très bref. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί πιστεύω ότι δυστυχώς και στην Επιτροπή μας αλλά και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάζεται το σχέδιο της Μόσχας με ένα θετικό τρόπο. Αυτό είναι μια προσωπική επίθεση λέει ο, ο βουλευτής χωρίς μικρόφωνο. Μα εγώ δεν μίλησα για κανένα, λέει ο κύριο Πρέντα. Κύριε Πρέντα, παρακαλώ συνεχίστε, λέει ο πρόεδρος. Εγώ δεν μίλησα για κανένα, προσωπικά, λέει ο κύριο Πρέντα. Εγώ θέλω να πω από τη δική μου πλευρά ο συνάδελφός μας ο Γκαμπριέλης Ραλτσπέργης δεν του επετράπει να μπει στη Ρωσία ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού μας Κοινοβουλίου για την ε, χώρα αυτή σε συνθήκες οι οποίες ήταν πραγματικά σαφείς ενώ είχε διπλωματικό διαβατήριο του είπαν ότι δεν μπορεί να μπει στο ρωσικό έδαφος και επομένως δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τους πολιτικούς του συνομιλητές κάτω από τέτοιες συνθήκες. Να έχουμε συναδέλφους οι οποίοι εκφράζουν τις απόψεις του Πούτιν και να μην ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα να μπουν οι συναδελφοί μας στη Ρωσία, αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο. <coughs> Κύριε Σαφχάουζεν, εάν θεωρείτε ότι σας αφορούν οι δηλώσεις του κύριου Πρέντα, σας δίνω τον λόγο. Να μην είμαστε υποκριτές κύριε Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι η παρέμβαση αυτή είχε αυτό το στόχο. Έχουμε μια σύγκρουση δύο μεγάλων δυνάμεων για τον έλεγχο της Ευρώπης μεταξύ άλλων αλλά και μεταξύ δύο οραμάτων κατά κάποιο τρόπο. Παρακαλώ θα ήθελα να πάρετε θέση για αυτό το οποίο είπε ο κύριο Πρέτα και όχι να αρχίσετε μια νέα παρέμβαση. Θέλω να πω ότι είναι πολύ εύκολο να λέμε ότι από τη μια πλευρά ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της Ρωσίας, ο πράκτορας της Ρωσίας. Μα εσείς μπορείτε να είστε με την ίδια λογική οι πράκτορες του, της Ουάσιγκτον. Αυτό είναι αναξιοπρεπές για το κοινοβούλιο μας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη βάση, την ιστορική βάση μιας σύγκρουσης η οποία μπορεί να μας οδηγήσει στον Τρίτο Παγκοσμίο Πόλεμο. Και σας λέω ξέρω γιατί μιλάω. Αγαπητοί συνάδελφοι. Γνωρίζουμε την κατάσταση της Ρωσίας. Πολλοί από εμά πήγαν εκεί πρόσφατοι, Η Ρεμπεκά Χάρμς, δεν μπόρεσε να μπει στη Ρωσία. Ζητήσαμε να αρθεί αυτή η απαγόρευση και το πράξαμε και στη συνέλευση των Πρόεδρων και όσο δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος για τον οποίο αυτό η ρωσική πλευρά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε ουσιαστικές σχέσεις με τη Ρωσία. Μας ε, είπε ο, ένας συνάδελφος ότι δεν μπόρεσε να μπει ο εισήτης ε, κύριος Λαντσπέρκης. Θα πρέπει να υπάρξει και μία επαφή με τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία για τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να γίνει αυτό στις 2 ή 3 Φεβρουαρίου. και επίσης ο κύριος Γκρόσμαν, ο πρόεδρος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου θα έρθει ενώπιον της Επιτροπής μας προς το τέλος του Φεβρουαρίου. Ενδεχομένως σε μια συνάντηση στο Στρασβούργο μπορούμε να προσκαλέσουμε τον κύριο Μπούσκοφ. Αν συμφωνείτε λοιπόν και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, μπορούμε να κάνουμε τις αντίστοιχες αυτές ε, προσκλήσεις. Ο κύριος Μπούσκοφ ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ρωσικής Δούμα θα μπορούσε ενδεχομένως να μας εξηγήσει την στάση της ε, Ρωσίας. Μπορούμε να το κάνουμε λοιπόν αυτό. Κύριε Σαφχάουζεν, μερικές φορές τα πράγματα είναι πολύπλοκα, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ σαφή. Η Ρωσία έχει περάσει τα σύνορα με μια γειτονική χώρα και έχει προκαλέσει πόλεμο στη γειτονική αυτή τη χώρα. Εμείς δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε αυτό. Έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο. Έχουμε ρωσικούς, ρω, ρωσικό στρατό στην Κρυμαία. Η Ρωσία έχει προσαρτήσει ένα τμήμα της Ουκρανίας και τώρα ασκεί πολεμικές ενέργειες στην Ανατολική Ουκρανία και έχει κάνει και αυτή την επίθεση στη Μαριούπολη. Όλα αυτά είναι γεγονότα. Τα γεγονότα δεν μπορούν να τίθενται υπό αμφισβήτηση. Και επομένως αυτή η πολιτική των ίσων αποστάσεων που αναφέρεται δεν μπορεί να ευσταθεί. Υπάρχει ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή εναντίον της Ουκρανίας και εμείς θα πρέπει μαζί με την ΟΑΣΕ να προστατεύσουμε το διεθνές δίκαιο και την Ουκρανία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει δεχτεί και η Ρουσία την ύπαρξη ενός διεθνούς δικαίου που δεν το έχει τηρήσει όμως. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την συζήτηση. Θα συνεχίσουμε εν ευθέτω χρόνο και επανεχόμαστε στην ημερήσια διάταξη. Είπατε και εσείς ε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για τον εκπρόσωπο της ε, των εξωτερικών υποθέσεων της Ράδα, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν είναι θέμα αποστάσεων, είναι θέματα ε, πολιτικής. Πρέπει να ακούσουμε και τους Ρώσους με τους οποίους διαφωνώ. Αλλά το να συνεχίσουμε να μιλάμε... Σας πρότεινα μόλις να καλέσουμε τον ε, επικεφαλής της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Δούμα, τον κύριο Πούσκοφ. Τη Δούμα. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι εννοούσατε του Ουκρανικού Κοινοβουλίου. Ο κύριο Πούσκοφ είναι ο πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Δούμα, λέει ο, ο κύριο Μπροκ. Okay, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Σημείο τη μέση διάταξη υπαριθμών 7. Αν μπορείτε να αναλάβετε την Προεδρία. Λοιπόν, επειδή έχουμε καθυστερήσει, να ξεκινήσουμε και να δώσω απευθεία το λόγο στον κύριο Παντζέρη. Ωραία. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Ησυχία παρακαλώ. Η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το 2013 βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι η εκπόνησή της ε, συμπίπτει με την ολοκλήρωση ε, του κύκλου, ο οποίος ξεκίνησε το 2012 από την Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Το στρατικό σχέδιο, το σχέδιο δράσης, των, ε, είπα το εκπρόσωπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, δράσεις τις οποίες ε, θα ε, ξαναξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος. Επομένως, η σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλη για μας. Οργανώσαμε μια σειρά από ακροάσεις, η πιο σημαντική ήταν το Νοέμβριο. Εκεί ακούσαμε όλους τους ενδιαφερομένους, Διακόπτει ο πρόεδρο. Ησυχία παρακαλώ. Αφήστε τον κύριο Παντζέρη να μιλήσει. Συνεχίστε παρακαλώ. Στην οποία ουσιαστικά συζητήσαμε με τις διάφορες ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις πώ θα πρέπει να συνταχθεί αυτή η έκθεση. Αποφασίστηκε να υπάρχει μία ε, ε θεματική προσέγγιση και όχι γεωγραφική ε, προσέγγιση και Υπάρχουν τρία, τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτή η επιλογή. Η πρώτη είναι πολιτική, γιατί το να συμπεριλάβουμε όλες τις χώρες του κόσμου σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε μια ένα η συζήτηση για το πώς ε, έχει κατάσταση στις διάφορες χώρες και να περάσει σε δεύτερο ε, επίπεδο ε, το πιο σημαντικό θέμα, πώς μπορεί να βελτιώσει την δράση προάσπισης και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Ο δεύτερος λόγος είναι πρακτικός. Η έκθεση ε, είναι ένα έγγραφο 372 σελίδων στην οποία συζητούνται πάνω από 150 χώρες. Αυτή είναι η έκθεση του Συμβουλίου. Εμείς πρέπει να περιλαμβάνουμε μία σαφή ε, σύνθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επομένως δεν έχουμε ούτε χώρο ούτε χρόνο να εξετάσουμε όλα τα θέματα ένα προς ένα. Και τρίτος λόγος, έχουμε την έκθεση του 2013 και είμαστε στο 2015 ήδη. Και είναι προφανές ότι έχουν υπάρξει αρκετέ αλλαγέ προ το χειρότερο και προ το καλύτερο, αλλά επειδή αναφερόμαστε στο 2013, είναι πιο λογικό να παραμείνουμε σε κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές αναθέμα και όχι γεωγραφικά. Πολύ σύντομα, ε, στη δομή της έκθεσης έχουμε την εισαγωγική ε, ενότητα που έχουμε τα διάφορα διεθνή ζητήματα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει ένα προήμιο το οποίο αναφέρεται ε, το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ένα πρώτο τμήμα στο οποίο γίνονται προτάσεις βελτίωσης των πολιτικών που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας. Ένα δεύτερο τμήμα το οποίο ε, αναφέρει διάφορα συγκεκριμένα μέσα τα οποία έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, υλοποίηση των ε, πολιτικών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα τρίτο τμήμα στο οποίο αναφέρονται συγκεκριμένε δράσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολυμερές επίπεδο και τρί, τέλος τα συμπεράσματα τα οποία αφορούν τη βελτίωση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προφανώς όλη αυτή η δουλειά ήταν αρκετά δύσκολη, διότι υποβλήθησαν περίπου 500 τροπολογίες και έχουμε συντάξει 25 συμβαστικές τροπολογίες. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια συνεδρίαση με τους πιο δυσυγητές, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω παρεπιπτόντων για την επικοδομητική συνεργασία και την ουσιαστική συνεισφορά στην ε, ε, σύνταξη αυτής της έκθεσης. Στην ε, συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν διάφορα κεφάλαια και καταλήξαμε σε συμφωνία για 25 συμβαστικές τροπολογίε και έγινε μια συζήτηση για κάποια σημεία επί των οποίων φυσικά θα ψηφίσουμε. Υπάρχει για παράδειγμα ένα θέμα το οποίο είναι πρόταση κάποιων ευρωβουλευτών να υπάρχει ένας ε, ειδικό εκπρόσωπος πλέον αυτού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο οποίος θα είναι υπεύθυνο για θέματα τα οποία σχετίζονται με τη διεθνή δικαιοσύνη και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Υπάρχει το θέμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω ενός μηχανισμού αναθεώρησης στις χώρες στις οποίες η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε αποτελέσματα. Μία συζήτηση για το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα έπρεπε να συντάξει ένα κατάλογο για του πολιτικού κρατουμένου παγκοσμίω και να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να συνδυάσουμε την ανάγκη να ε, εξετάσουμε τι διάφορε περιπτώσει συστηματικά χωρί να αποτελεί αυτό κίνδυνο για του ανθρώπου που προσπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικά υπάρχουν και κάποια προβλήματα, θέματα τα οποία αντιμετωπίσαμε, στα οποία πρέπει να βρούμε μια μέση λύση ή θα πρέπει να ψηφιστούν και αφορούν συγκεκριμένε γεωγραφικέ περιοχέ, κυρίω ε, Μέση Ανατολή και Δυτική Σαχάρα. Υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία υπάρχει σημαντική επιβεβαίωση και καινοτομία στην έκθεση. Αναφέρομαι για παράδειγμα στο θέμα των ανηλίκων και να σας αναφέρω μόνο γιατί δεν υπάρχει χρόνος να τα συζητήσουμε όλα. Ε, άτομα με αναπηρία, ε, θρησκευτικέ το πολύ σημαντικό θέμα της βίας κατά των γυναικών, ε, πολιτικός γάμος μεταξύ ομοφύλων. Ε, κατάργηση της θανατικής ποινής ε, και των βασανισμών και αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου όσον αφορά το θέμα των συνόρων, γεγονός που παρακολεί τη δυνατότητα των μεταναστών να κάνουν αίτηση ασύλου. Υπάρχει σημαντική ε, νομική αναγνώριση για το καθεστώς του κλιματικού πρόσφυγα και τέλος υπάρχει και το θέμα των νέων προσανατολισμών για τις ε, κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες ε, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία από τη διάσκεψη των Πρόεδρων των Αντιπροσωπιών ε, με τον πρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, έχουμε γνωμοδότηση από τις Επιτροπές ε, ΔΕΒΕ και ΛΥΜΠΕ. Οι τροπολογίες που προτάθηκαν από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τα δικαιώματα των γυναικών και των ε, ε, κοριτσιών καλύπτονται ήδη από την έκθεση, αλλά θα τα λάβουμε και αυτά υπόψη. Όσον αφορά την Επιτροπή ανάπτυξη, η Επιτροπή Ανάπτυξης συνεισέφερε ουσιαστικά και εγώ έβαλα ένα ειδικό κεφάλαιο για τα θέματα των παιδιών με αναπηρία και υπάρχει ειδικό κεφάλαιο γι' αυτό και συγκεκριμένε τροπολογίε και υπάρχουν και κάποιε ενδιαφέρουσε προτάσει που προέκυψαν από διάφορε πολιτικέ ομάδε, των Πρασίνων για παράδειγμα, και φτιάξαμε και δύο κεφάλαια. Ένα για τη σχέση αθλητική δραστηριότητα και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, ένα κεφάλαιο για τα ναρκωτικά και θα υπάρχει και μια προφορική ε, ε, τροπολογία από πλευρά μου. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μας οδηγούν στην ε, πολύ σημαντική ε, συνεισφορά που έχουν στην ε, ζωή των ανθρώπων και θα πρέπει να αποτελέσουν βάση για τα θεμελιώδεις ανάγκες και την αξιοπρέπεια του κάθε ατόμου. Γι' αυτό ακριβώς και ήθελα ευθύ εξ αρχής ε, να είμαι πιο διάφανο και να προσπαθήσω να συμπεριλάβω όσο περισσότερα γίνεται και επ' αυτή τη βάση και βάσει και τη καλή συνεργασία με όλου του και οδησηγητές του οποίους και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω, ελπίζω ότι η έκθεση θα μπορέσει να λάβει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη στην ψηφοφορία που προβλέπεται για τι 9 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο ε, για την Επιτροπή μα. Τελείωσα. Ο κύριος Πρέντα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Παντζέρη για είδαμε γύρω από τις, ε, ε, ήδη τις συμβεβαστικές τροπολογίες συναντηθήκαμε με τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους ε, συζητήσαμε γύρω στις 28 συμβιβαστικές ε, μετά από προτάσεις του εισηγητή και από την άποψη του ΕΛΚΑ εγώ στους κοιόδους εισηγητής συμφώνησα με 19 συμβιβαστικές από τις 28 θα επανέλθουμε σε αυτές και το, το, το, η θέση που στήριξα οι θέσεις μάλλον που στήριξα σχετίζονται με τροπολογίες που μας επιτρέπουν καλύτερα να λάβουμε υπόψη την υπόθεση της δημοκρατίας, διότι Γιατί το είπα ήδη σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση, το κείμενο που θα ψηφίσουμε αφορά τόσο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσο και για τη δημοκρατία. Και γι' αυτό επέμεινα να αναφερθεί και να υπάρχει και μια δημοκρατική μνήμα. Μέσα στο πλαίσιο αυτών των ε, τροπολογιών επαναλάβαμε την σταθερή μας στήριξη για την ύπαρξη ενός προσώπου της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω πως συμφωνούμε με τους πράσινους και επιμένω ιδιαίτερα για το γεγονός ότι πρέπει να χαιρετήσουμε το εξαίρετο έργο τον, ε, του εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης εκφράσαμε με τους φιλελεύθερους συνάδελφους την επιθυμία μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί από ό,τι μέχρι τώρα. Γενικότερα με τους συνάδελφους σοσιαλιστές, τους φιλελεύθερους, τους πράσινους αλλά και το FDD ε, συμφωνήσαμε για τη σημασία της απόρριψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο όλων αυτών των ε, θεμάτων. Επίσης συμφωνήσαμε με τους πράσινους συνάδελφους και στους σοσιαλιστές για τη σημασία της προστασίας του παιδιού, ιδιαίτερα σε περιστάσεις πολέμου, σε κατάσταση πολέμου. Αλλά είχαμε και ε, διάφορα σημεία που δεν συμφωνήσαμε και ως σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚΑ χρειάστηκε να αρνηθώ κάποιες ε, συμβιβαστικές που προτάθηκαν. Όπως η συμβιβαστική 26 που, που μιλούσε για τη μετανάστευση και για τη μεταρρύθμιση της ε, συνθήκης του Δουβλίνου. Πιστεύουμε όμως εμείς ότι ένα τέτοιο θέμα πρέπει να συζητηθεί στη ΛΥΜΠΕ. Δεν πρέπει να εμείς να αντικαταστήσουμε τους συναδέλφους μας της ΛΥΜΠΕ. Και αυτό είναι και το επιχείρημα που πρότεινα. Στη συνέχεια αποσυρθήκαμε από την ε, ε, συμβιβαστική 10 που ζητούσε να εκφραστεί για το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες με γενικό τρόπο. Εγώ θεώρησα ότι το να αναφερθούν οι καλές προθέσεις και η πραγματική δέσμευση μπορεί να είναι πολύ προβληματικό. Διότι δεν μπορούμε αυτό να το μετρήσουμε. Και γι' αυτό αρνηθήκαμε να συνυπογράψουμε την 10 γενικότερα και εδώ απλά δίνω το παράδειγμα της Συμβαστικής 18 αρνήθηκα τις ψευδοσυμβιβαστικές όπου, όπου χρησιμοποιούνται λέξεις που είναι περιθωριακές δεν είναι καθόλου ουσιαστική σημασία σε μια συμβιβαστική που αφορά ένα πολύ λεπτό ζήτημα, αλλά όπου η θέση του ΕΛΚΑ δεν εκπροσωπείται τελικά καθόλου. Εδώ την αρνήθηκα λοιπόν τελείως αυτή τη συμβιβαστική. Όσον αφορά τις ε, τροπολογίες που πρότειναν οι συνάδελφοι του ΕΛΚΑ, προσπάθησα να μείνω πιστός στο πνεύμα αυτών Οπότε στήριξα και ζήτησα και από τον εισηγητή να διατηρήσει τις τροπολογίες που πρότειναν οι συνάδελφοι αντί να εισάγουμε λανθασμένα κατά κάποιο τρόπο ή αυτές τις τροπολογίες σε συνδεστικά κείμενα. Τέλος, να συμπώ ότι δεν συμφωνούμε καθόλου για την επανεισαγωγή ακόμα μια φορά του θέματος της Δυτικής Σαχάρας ως ε, σημείο αυτής της έκθεσης. Το να μετατρέψουμε τη Δυτική Σαχάρα στο πιο σημαντικό σημείο αυτής της έκθεσης είναι απαράδεκτο. Υπάρχουν πολλά άλλα μέρη όπου τίθεται όπου υπάρχουν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το να κάνουμε μια τροπολογία και να αναφέρουμε μόνο τη Δυτική Σαχάρα δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί κατά τα άλλα είναι εξαίρετη η έκθεση η, η έκθεση του κυρίου Τάνοκ που έφτιαξε πέρσι για το Σαχέλ δεν μιλούσε για τη Δυτική Σαχάρα και τελικά μετά από τεράστιες πιέσεις, αντί να μιλάμε για το Σαχέλ, μιλήσαμε για τη Δυτική Σαχάρα. Αυτή η τόσο σημαντική έκθεση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία θα ήταν άπρεπο να μετατραπεί σε μια υπόθεση για τη Δυτική Σαχάρα. Υπάρχουν ένα σωρό φρικτές υποθέσεις στον κόσμο. Αυτές δεν αναφέρονται καθόλου και ενώ γίνεται απόπειρα να περάσει αυτό το θέμα και θα χάσουμε τη συζήτηση στην Ολομέλα. Θα είμαστε εκτός θέματος άμα επικεντρώσουμε την προσοχή μας εδώ. Υπάρχουν ε, σχεδόν 500 τροπολογίες από συναδέλφους που ντε και καλά θέλουν να περάσει αυτό το θέμα. Εγώ νομίζω πως δεν πρέπει να δεχτούμε ούτε μια αναφορά σε ένα μέρος στην έκθεση αυτή. Γιατί όπως είπε και ο κ. Παντζέρη συμφωνήσαμε για τα θέματα και συμφωνήσαμε και για να γίνει ένας πλήρης κατάλογος για όλες τις υποθέσεις που συζητάμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλες τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν δεν μπορώ να δεχτώ ότι αντί να συζητάμε για αυτή την γενική κατάσταση που αφορά όλες τις χώρες και ε, να αντικαταστήσουμε με την ε, Δυτική Σαχάρα, λες και αυτό είναι το μόνο θέμα. Έχουμε άλλες ευκαιρίες και άλλα μέρη για να συζητήσουμε. Αυτό το μέρος του κόσμου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο κύριος Χάουιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Παντσέρη για την πολύ καλή έκθεσή του. Νομίζω ότι έχει κάνει σωστές επιλογές, έχει παραμείνει στον θεματικό τρόπο παρουσίασης και όχι να έχει μια προσέγγιση που να εστιάζει σε συγκεκριμένες χώρες. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Πρέντε για τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά νομίζω ότι η προσέγγιση θα πρέπει να είναι ουδέτερη σε σχέση με τις χώρες, θα πρέπει να έχει θεματικό χαρακτήρα και πρέπει να εξασφαλίσουμε στην τελική ψηφοφορία ότι θα υποστηρίξουμε την προσέγγιση του εισηγητή. Εγώ θέλω να υποστηρίξω ιδιαίτερα αυτά που λέει ο κύριος Παντσέρη για τα δικαιώματα τα εργασιακού χαρακτήρα. Στην εξαγωγή των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων και αυτά που λέει τώρα για τη βία μετά από τις αποφάσεις που πήραμε πέρσι για το βραβείο Σαχάρο και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παράγραφος 52 σε σχέση με την ε, προστασία των ομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παίρνουν μια χρηματοδότηση. Εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε τις ομάδες αυτές και τη διατύπωση στην παράγραφο 52. Οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 24 ξέρουμε ότι κάποιες αντιπροσωπείες σε παγκόσμιο επίπεδο δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα αυτό και κάποιες είναι πιο αποτελεσματικές από τις άλλες να παρακολουθούν τις δικαστικές διαδικασίες, να επισκέπτονται αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη φυλακή αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει όχι μόνο η δημόσια διπλωματία, αλλά να υπάρξουν και οι απαραίτητε ενέργειε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ιδιωτικό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι σωστή η ισορροπία που επιτυχάνει ο κύριο Παντσέρη. Βλέπω ότι λέει στην έκθεσή του πρέπει να υπάρχει και μια έκθεση για την υλοποίηση όλων αυτών με στόχο να μπορούμε να έχουμε κάτι το ουσιαστικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην παράγραφο 44 τονίζει ότι υπάρχει μια ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι τα θύματα της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν υποστεί παραβίαση των δικαιωμάτων τους από επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα προσφυγής. Και εγώ ήμουν παρόν στην ε, συνδιάσκεψη της Γενέβης που αφορούσε δεσμευτικού χαρακτήρα εργαλεία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι μια συζήτηση με τα κράτη-μέρη για το θέμα αυτό θα μπορούσε να τεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ολομέλεια. Και σε σχέση με την σύμβαση για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες ε, φέτος θα έχουμε την πρώτη έκθεση παρακολούθησης για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να είναι τμήμα της συζήτησης, όχι μόνο στην Επιτροπή μας, αλλά και στην Ολομέλη, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα έτη τα οποία θα ακολουθήσουν. Είναι πολύ καλή έκθεση και θέλω να συγχαρώ τον κύριο Παντσέρη για αυτήν. Ελπίζω λοιπόν θα έχει μεγάλη υποστήριξη και στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου μας. Ο κύριος Τάνοκ. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Παντσέρη, εξ ονόματος της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ο κύριο Χένκελ δεν μπορούσε να είναι παρόν μαζί μας. Απόψε θέλω να πω έσμενα λόγια εξ ονόματός του και εξ ονόματος της ομάδας μας. Έχει καταθέσει 14 τροπολογίες κύριο Χένκελ. Θα γνωρίζουν οι συνάδελφοι ποια είναι τα κύρια θέματα τα οποία τον απασχολούν. Εγώ έχω παρακολουθήσει πολλά χρόνια τις αιτήσει εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια εποχή ο Ρίτσαρτ Χάουερτ και εγώ ήμασταν αντιπρόεδροι της Επιτροπής, Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό το οποίο τονίζει η ομάδα μου κάθε χρόνο είναι ότι δεν πρέπει να λοξοδρομήσουμε και να βγούμε από τον χώρο των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μπούμε στον χώρο των κοινωνικών δικαιωμάτων που εκεί εισέρχονται ιδεολογικές αξίες που προέρχονται από άλλες πολιτικές ομάδες. Και εμείς λοιπόν έχουμε κάποιες ανησυχίες για κάποιες πτυχές της έκθεσης, όπως η επιχείρηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι τέσσερις παραγράφοι που ακολουθούν, ή παράγραφος 76 για την αρπαγή γης. Αυτά είναι προτεραιότητες δεύτερης κατηγορίας τη στιγμή που σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως οι ISIS που εκτελούν και αποκεφαλίζουν αθώους ανθρώπους, χριστιανούς, Ιεζιντοί, ε, Σιήτες, πουλάνε γυναίκες σαν σκλάβες. Μια βαρβαρική πρακτική από, τη, από το Μεσαίωνα. Εκεί λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, όχι θέματα οικονομικού χαρακτήρα. Και η ομάδα μου δεν έχει κάποια συλλογική άποψη για τα θέματα αυτά. Θεωρεί ότι θέματα όπως ε, τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα είναι θέμα ατομικής συνείδησης. Τα θέματα της, ε, του Συμφώνου Συμβίωσης ή των γάμων ατόμων του ίδιου φύλου δεν θέλουμε να έχουμε μια κοινή στάση στα θέματα αυτά. Κατανοούμε όμως ότι είναι ζητήματα όπου ο καθένας θα πρέπει να ακολουθήσει την προσωπική του συνείδηση. Ευχαριστώ ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι φιλελεύθεροι συμμετείχαν ε, ενεργά στη συζήτηση και έδωσαν μάχη για το συμβιβαστικό κείμενο. Ε, προτείναμε 13 τροπολογίες ε, στο κείμενο και να συγχαρούμε και τον κύριο Παντζέρη, ο οποίος από πλευράς μου θεωρώ ότι δημιούργησε πολύ θετικό κλίμα και προσπάθησε να εξεύρει την καλύτερη δυνατή συμβαστική λύση. Και δεν πήρε η κάθε πολιτική ομάδα το συμβιβασμό που αναζητούσε βέβαια, αλλά αν δούμε τα βασικά τμήματα του κειμένου που έχουμε μπροστά μας, θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με το κείμενο. Οι φιλελεύθεροι ε, έχουν συμφωνήσει σε εννέα τροπολογίες και θεωρώ ότι το κείμενο αντανακλά και αναγνωρίζει πολύ συγκεκριμένε τάσεις ε, στην πολιτική μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες. Η έκθεση είναι πιο εξορθολογισμένη και η ποιότητα της έκθεσης αυτής έχει βελτιωθεί κατά την άποψή μου αν τη συγκρίνουμε με τις εκθέσεις των προηγούμενων ετών. Περιμένουμε με ανυπομονωσία και την έκθεση για το 2014. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε και τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε και να αναλύσουμε κάποιες νέες τάσεις ε, στην πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως όσον αφορά επιθετικές πολιτικές από κάποιες γειτονικέ χώρες, για παράδειγμα ε, την Ουκρανία, ε, προς την Ουκρανία μάλλον. Και φυσικά θα ήθελα να υπάρχει μια ισχυρή γραμμή πολιτικής για την επόμενη έκθεση για το 2014. Κύριε Πρόεδρε, για να συνοψίσω, νομίζω ότι δικαίως πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με τη συμβαστική έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας και ε, προσβλέπω στην τελική ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λοχπίερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή και για το σχέδιο κειμένου αλλά και ε, για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Εμείς συμμετέχουμε σε 8 συμβιβαστικές λύσεις και κάνατε πολύ καλή δουλειά, σε 18 συγγνώμη. Ε, υπάρχουν κάποια καλά σχόλια και γραπτές προτάσεις ε, για το σχέδιο των συμβιβαστικών τροπολογιών και όπως είπατε έχετε και εσείς μια προφορική τροπολογία για τους απάτριδες. Όσον αφορά τις ε, τροπολογίες μας, έχουμε υποβάλει αρκετές για την ενίσχυση των ανθρώπων που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως ε, αυτούς που δίνουν μάχη για οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, συνδικαλιστικά ε, σωματεία και θέματα αρπαγής γης. Είναι θέματα τα οποία έχουν προκύψει και από τη γνωμοδότηση της ΔΕΒΕ για τις ε, διαδικασίες αρπαγής γης ε, υπάρχουν ε, κάποιοι ακτιβιστές που ασχολούνται με το θέμα και έχουμε μία παράγραφο που προτείνουμε για να αντιμετωπίζουμε αυτές τις περιπτώσεις. Για τους ανθρώπους που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα επισημαίνουμε το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζει ή να επεκτεί, στον ίδιο βαθμό ή να επεκτείνει τη χρηματοδότηση για τα θέματα αυτά. Όπως είπε και ο εισηγητής και ο κύριος Πρέντα για τον ειδικό εκπρόσωπο για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, εμείς είμαστε υπέρ μιας ξεχωριστής θέσης και αυτό σε καμία περίπτωση δεν ε, ε, υπονομεύει το έργο του ειδικού εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί κάνει καλή δουλειά και έχει πολλή δουλειά να κάνει. Αλλά θεωρούμε και έχουμε συμφωνήσει και σε προηγούμενη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι ένα ειδικό εκπρόσωπο για το ανθρωπιστικό διεθνέ δίκαιο είναι πολύ σημαντικό ε, ρόλο και θα πρέπει να ενισχύσει και την παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολυμερή βήματα για το θέμα αυτό. Επίσης έχουμε μια ειδική παράγραφο για την ε, ε, εμπορία ανθρώπων και το γεγονός ότι θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Και έχουμε μια παράγραφο για τον αθλητισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, στην προηγούμενη συζήτηση για την Ουκρανία αναφέρθηκε ότι θα γίνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Ρωσία. Έχουμε και ευρωπαϊκούς αγώνες φέτος και θα πρέπει να συζητήσουμε και με αθλητικές ομοσπονδίες και με όσους διοργανώνουν τέτοιες αθλητικές εκδηλώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Επίσης θέλουμε ε, ε, και μία παράγραφο για τα drones ε, βάσει και τα νόσα είχαμε στο ψήφισμα του Φεβρουαρίου του 2014. Έχουμε κάποιες ακόμα τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι θα καθυστερήσουμε πολύ τώρα να τις αναφέρω μία προς μία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοράου. Va bene, abbiamo... Grazie. Μιλήσαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όντω το κείμενο του εισηγητή Μπαντζέρη είναι καλό συμβαστικό κείμενο. Παρατηρήσει ε, δε τη κυρία Λοχομπίλερ με βρίσκουν σύμφωνα θα λοιπόν, και εμείς είμαστε υπέρ για ένα δεύτερο μια δεύτερη μορφή αντιπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Bueno, ahora me toca a mí. Nosotros no Λαμβάνω και εγώ το λόγο. Εμείς δεν συμμεριζόμαστε την ε, γενική κατεύθυνση αυτής της έκθεσης η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δίνει διδάγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Δεν θέλουμε μια παρεμβατική αντιμετώπιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ούτε μας αρέσει το να αντιγράφουμε τις πρακτικές των Ηνωμένων Πολιτειών όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Γι' αυτό το λόγο έχω καταθέσει πολλές τροπολογίες, σχεδόν 28, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία λείπουν, η κατάσταση του λαού της Παλαιστίνης, οι εξαφανισμένοι του Μεξικού, αυτοί οι οποίοι έχουν οι δεκατούμενοι στο Γουαντάνο της ΗΠΑ και η σύγκρουση στην Δυτική Σαχάρα. Το Κοινοβούλιο όμως έχει, το δικαίωμα, έχει το, την υποχρέωση να καταδικάσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Μαρόκο εναντίον του λαού των Σαχαραουή στα κατεχόμενα δάση Σαχάρας. Δεν ναι, συμφωνώ με τον κύριο Πρέντα ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκδιώχθησαν όταν προσπάθησαν να μπουν στην Δυτική Σαχάρα. Και το Κοινοβούλιο έχει εκρεμή ε, αποστολή για να πάει στη κατεχόμενη Δυτική Σαχάρα και του να δει τους κρατούμενου του Σαχαραούι που δεν έχει λειτουργήσει γιατί το εμποδίσει το Μαρόκο. Στη χώρα μου είναι ένα καυτό θέμα. Ο Χασάν Άλια έχει αντιμετωπιστεί με σκανδαλώδη τρόπο από την Υπουργείο Εσωτερικών της χώρα μου. Γιατί δεν του έδωσε την δυνατότητα να πάρει άσυλο ενώ έχει καταδικαστεί σε ισόβια δεσμά από τι κατοχικέ δυνάμει στη Δυτική Σάχαρα. Η Μινούσο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ε, περιοχή της Δυτικής Σαχάρας δεν έχει κάνει τίποτα για να επιταχύνει το δημοψήφισμα στην περιοχή αυτή και την απελευθέρωση των ε, κρατουμένων στις ε, φυλακές του Μαρόκου. Ελπίζουμε ότι ο ΣΥΤΙΣ θα λάβει υπόψη το παγκόσμιο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα Ηνωμένα Έθνη. Εμείς δεν πρέπει να ακολουθούμε την ατζέντα του Μαρόκου και δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι μόνο το Μαρόκο και η Αλγερία παίζει σε αυτό το παιχνίδι, τη στιγμή που είναι σαφέ από άποψη διεθνούς δικαίου ότι το μέτωπο Πολυσάριο είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του λαού των Σαχαραουή. Το Μαρόκο λοιπόν είναι αυτός ο οποίος κατέχει τη Δυτική Σαχάρα σε βάρος των Σαχαραουή. Δεν υπάρχουν άλλοι οι οποίοι εμπλέκονται και δεν θα είμαστε συνένοχοι τη χειραγώγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με αυστηρότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα πάντα τα οποία μπλέκονται και το διεθνέ δίκαιο. Ο κύριο Μίλιαν Μόν έχει το λόγο. Εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή και πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια θεματική προσέγγιση. Αυτή πρέπει να είναι η γραμμή που ακολούθησε ο κύριο Πρέντα και τον υποστηρίζω. Και ο κύριο Χάουιτ, ο συντονιστή των Σοσιαλιστών. Κατέθεσα και εγώ κάποιες τροπολογίες σύντομες που πήγαν προς αυτήν την κατεύθυνση για μια θεματική έκθεση. Πρέπει να είμαστε λοιπόν συνεπείς. Αν ο εισηγητής θέλει να έχει μια θεματική προσέγγιση, είναι δύσκολο και μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες να αναφέρουμε γεωγραφικά προβλήματα. Αν κάτσουμε και καταλογραφήσουμε όλες τις χώρες όπου υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι πολλές αυτές οι χώρες, μέσα στο πλανήτη μας. Η εκθεσή μας θα θεωρηθεί ότι είναι διακριτικού χαρακτήρα, ότι έχει μεροληπτικό χαρακτήρα, ότι δίνει έμφαση σε ορισμένου τομεί και όχι σε άλλου. Και εγώ θέλω να παρακινήσω λοιπόν τον εισηγητή να είναι συνεκτικός με την αρχική του προσέγγιση για μια θεματική προσέγγιση. Αλλιώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να κάνει η εκθεσή μου για ένα θέμα τόσο ευαίσθητο και τόσο σημαντικό στα ανθρώπινα δικαιώματα να, να εστιάσει σε τρεις ή τέσσερις καταστάσεις χωρών. Αυτό θα της αφαιρέσει την ισορροπία και την απαραίτητη απόσταση που πρέπει να έχουμε και τόνισε ο εισηγητής ότι η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι θεματική προσέγγιση. Η κυρία Γκάμισ. Εγώ πιστεύω πως είναι σημαντικό να έχουμε εδώ την αιτήσια για τα ανθρώπινα δικαιώματα ένα λόγο, γιατί είναι ένας τρόπος για να θυμίσουμε στις κυβερνήσεις μας ότι πρέπει να είναι συνεπείς και συνεκτικές στην προσέγγιση τους στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως τα έπρεπε και στις εσωτερικές τους πολιτικές. Κατανοώ την προσπάθεια και ευχαριστώ πολύ τον ε, τον Παντζέρη για τη δουλειά του που αποτελεί εξαιρετική βάση αλλά και τη δουλειά και την προσπάθεια που έκανε για να μπορέσει να χωρέσει και όλες τις τροπολογίες ε, που κατέθεσαν οι συνάδελφοι όπως και εγώ ίδια και καταλαβαίνω και την προσπάθεια για εξορθολογισμό ε, των διαφόρων ομάδων. Αλλά δεν πιστεύω πως η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να να είναι, πώς το λέμε, πώς το λέμε, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένες καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ως προς αυτό, και ήμουν μία από τον όσων επέβαλα ανθρωπολογίες για τη Δυτική Σαχάρα, και αυτό διότι ε, πρόκειται για, μια, για ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο δεν είναι μόνο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά σαφώ είναι και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θέλω να πιστήσω ε, η προσοχή σα στο γεγονό ότι το πρώτο άρθρο του Διεθνού Συμβούλου για τα πολιτικά και, ε, ε, και πολιτιστικά δικαιώματα είναι ακριβώς το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Είναι το πρώτο άρθρο το βασικό νόμο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα των λαών είναι αυτά που παραβιάζονται και λόγω αυτών στη συνέχεια παραβιάζονται και δεν εξασφαλίζονται και τα ατομικά δικαιώματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είμαστε φίλοι του Μαρόκου, αλλά δεν θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να ακολουθήσουμε διδακτική της Τρουθοκαμίλου. να κρύβουμε το θέμα. Το Μαρόκο πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα στο πλαίσιο του ΙΕ και δεν δέχομαι τη θέση των κρατών μελών μας που απλώς ε, δεν το φύγουν για να μην τεκωθούν με τους φίλους μας στο Μαρόκο. Τελείωσε ασυνεπή θέση. Όχι μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και για το διεθνέ δίκαιο. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο θέλω να αναφερθεί η Δυτική Σαχάρα. Μα δεν υπάρχει πουθενά κατάλληλο χώρο για να ε, μιλήσουμε για αυτό το θέμα και το ξέρω πάρα πολύ καλό εδώ, γιατί ε, είμαι χρόνια εδώ. Ποιε δυσκολίε είχαμε να επισκεφθούμε τη Δυτική Σαχάρα και τι φυλακέ. Και εγώ ήμουν μέρο τη αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε τη Δυτική Σαχάρα όχι κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, μια αντιπροσωπεία της ομάδας μου και προσπαθήσαμε να επισκεφθούμε τους ε, ε, κρατούμενους στις φυλακές της Ραμπάτ και δεν μας άφησαν. Δεν μπορέσαμε ούτε καν επισκεφθήκαμε την φυλακή του Λαγιούν, αλλά δεν μπορέσαμε να συνομιλήσουμε με τους κρατούμενους, πράγμα το οποίο είναι τελείως απαράδεκτο. Δεν είναι καλή πολιτική λοιπόν όσων λένε ότι είναι φίλοι του Μαρόκου να συνεχίσουν να κάνουν τα στραβά μάτια. Και επίση, εμεί μιλάμε και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι σωστό να αναφερθεί και εν πάση περιπτώσει, όσοι έχουμε υποβάλει αυτή την τροπολογία δεν το καταλήγουμε και κάθε ομάδα θα αναλάβει τις ευθύνε της. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τα στραβά μάτια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Δυτική Σαχάρα που βεβαίω συνδέεται με το θέμα της αυτοδιάθεσης για τον λαό της Δυτικής Σαχάρα. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες και τώρα το λόγο έχει ο Ρικάρδο Σέρι από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εμείς από πλευράς μας υποστηρίζουμε στεναρά αυτή την έκθεση διότι θεωρούμε ότι έχει επικεντρωθεί στα συγκεκριμένα θέματα και επίσης χαιρόμαστε και για την προσέγγιση που έχει ακολουθήσει ο κύριος Παντζέρη ε, σε αυτή την έκθεση με τις θεματικές ενότητες. Όπως είπε και ο κύριος Παντζέρη, η έκθεση αυτή είναι πολύ επίκαιρη διότι έρχεται στο τέλος αφενός της εφαρμογής ε, του παρόντος προγράμματος δράσης για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αρχή της διαδικασίας ε, συζήτησης ενός νέου σχεδίου δράσης και πρότασης κάποιων νέων δραστηριοτήτων για το μέλλον. Θεωρούμε λοιπόν ότι η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και πολύτιμη ε, γιατί κάνει πολύ συγκεκριμένε προτάσεις και φυσικά θα τις λάβουμε υπόψη. Κάποια από τα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω είναι ε, σίγουρα ο κεντρικός ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πολιτική μας εν γέννη η πολύ σημαντική προσοχή στον εξορθολογισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε όλα τα ζητήματα, κάτι το οποίο κάναμε και στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα στην εφαρμογή του νέου σχεδίου δράση και ίσω είναι και η βασική μα προτεραιότητα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά επίση θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμα κάποια από τα ε, συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία προτείνονται στην έκθεση, κυρίω όσον αφορά τη συγκεκριμένη εφαρμογή των μέσων μα. Έχουμε μία σειρά από μέσα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εφαρμόσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα επιτόπου. Πρέπει να βελτιώσουμε αυτά τα μέσα, πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα εφαρμόζουμε και ε, υπάρχουν χρήσιμε προτάσει από την έκθεση. Κάποιε από αυτέ τι προτάσει αναφέρθηκαν, κάποια από αυτά τα μέσα αναφέρθηκαν, για παράδειγμα διάλογοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβάνονται και το ρόλο των αντιπροσωπείων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να βελτιώσουμε τα μέσα αυτά και βεβαίως αυτό θα γίνει σε ε, ε, συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον. Νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ και επίση θα πρέπει να σα ενημερώσω πολύ σύντομα ότι ετοιμάζουμε την ετήσια έκθεση, μια νέα ετήσια έκθεση που θα καλύπτει το 2014, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι έτοιμη για τον Ιούνιο φέτο και φυσικά προσβλέπουμε και στην εφαρμογή της δικής σας της έκθεσης, της έκθεσης Παντζέρη στους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή. Κύριε Παντζέρη. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους τις εισηγητές που πανέλθαν. Ευχαριστώ τον κύριο Χάουετ για τα καλά του λόγια. Νομίζω πως στην ουσία ισχύουν οι προϋποθέσεις για να κάνουμε μια καλή δουλειά και ελπίζω πως όντως θα γίνει αυτό. Θα σταθώ μόνο σε δύο σημεία. Το πρώτο αφορά τη Δυτική Σαχάρα. Εγώ επειδή ε, Θεώρησα ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να βασιστεί στα θεματικά ζητήματα. Συμφωνώ με τον Πρέντα που λέει ότι δεν ήταν σκόπιμο να σταθούμε σε γεωγραφικά ζητήματα. Ωστόσο, έλαβα μια εντολή από πλευρά των σχεδόν εισηγητών για το γεγονός ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μια ε, υπόθεση όσον αφορά την, μια συμβαστική λύση. Ε, έφτασαν κάποιες προτάσεις, το λέω άμεσα. Εάν δεν μπορέσουμε λοιπόν να βρούμε συνδεστική για αυτό το θέμα, η γνώμη μου είναι να είμαστε αρνητικοί για όλες τις τροπολογίες που υπευλήθησαν, διότι βεβαίως εάν επανέλθουμε στην αρχική θέση, ε, η θέση αρχική ήταν να μείνουμε στο θεματικό πεδίο. Εγώ δεν θέλω να πω με αυτό ότι όχι, δεν θέλω ούτε και να το ξαναπώ. Ότι αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, οκ, αδιαφορετικά επανερχόμαστε στην πρώτη βάση εργασίας που ήταν ε, τα, ε, η θεματική. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση του ειδικού απεσταλμένου για το διεθνές δίκαιο, κατανοώ τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις, η γνώμη μου είναι κάπως διαφορετική, διότι ε, θέλει να επεκτείνει την εντολή του ειδικού απεσταλμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και εδώ θα πρέπει η δημοκρατία να αποφασίσει για τις ε, τροπολογίες, οπότε θα το ψηφίσουμε. Θα ψηφίσω αν περάσει αυτό και διαφορετικά σημαίνει ότι ε, απλώς παρατείνεται η εντολή στον ε, τωρινό εκπρόσωπο. Αυτά έχω να πω και ελπίζω ότι στις 9 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε με μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων υπέρ αυτής της έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παντσάρη. Έχουμε κλείσει αυτό το σημείο. Στις 9 Φεβρουαρίου θα είναι η επόμενη μας συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Συνεδριάσουμε πρώτα στις 2 Φεβρουαρίου στις 3 η ώρα. Και τώρα θα αρχίσει η συνεδρίαση του Διευρυμένου Προεδρείου. Διακόπτω για 5 λεπτά.